Euh, Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας πρότεινα να ξεκινήσουμε μέσω τη εργασίες μας. Το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η υιοθέτησή της. Υποθέτω πως δεν υπάρχουν κάποιες προτάσεις ή σχόλια. Εγκρίνεται λοιπόν. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η ειδική μας ε, η Επιτροπή μας, η Ειδική Επιτροπή μας, έχει σήμερα μια έκτακτη συνεδρίαση στην οποία θα έχουμε δύο πολύ σημαντικά, δύο σημαντικές ακροάσεις. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε τους μετά τους επιτρόπους μάλλον, Μοσκοβισή και Φερστάγκερ. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με την Προεδρία του Λουξεμβούργου Και μετά τις 6 ώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεις, απόψεων με τέσσερις ε, υπουργούς οικονομικών από ε, χώρες της Ένωσης. Χαίρομαι λοιπόν για αυτό το πνεύμα συνεργασίας που έχει επιδείξει το Συμβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω πρώτα απ' όλα δύο ομάδες επισκεπτών που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σε αυτή τη μικρή κατά τα λάθουσα. Πέρα από τους εκπροσώπους του τύπου που παρευρίσκονται στην δική μας ειδική επιτροπή τάξη όπως και σε πολλές άλλες επιτροπές ε, του Κοινοβουλίου, τον οποίων οι συνεδριάσεις εξάλλου μεταδίδονται και με web streaming στο διαδίκτυο. Έχουμε λοιπόν μια ομάδα από τη Σαξονία της Γερμανίας, από το τοπικό κοινοβούλιο, από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και επίσης ε, μια ομάδα από το, ε, μαθητών από το Γιβραλτάρ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω επίσης τα μέλη της Επιτροπής ΤΑΞ ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στην έκθεση έχει παραταθεί κατά 24 ώρες και λήγει αύριο στις 2 το μεσημέρι. Δόθηκε αυτή η παράταση για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να λάβετε υπόψη τις απαντήσεις που θα ακούσουμε απόψε. Θα σας ενημερώσω επίσης ότι ότι είχαμε αποστείλει αντιπροσωπείες ορισμένες χώρες, μία από τις οποίες ήταν το Λουξεμβούργο. Και σας ευχαριστώ για αυτό κύριε Υπουργέ. Για την υποδοχή που τους επιφυλάξατε και εσείς και η Δημόσια Δίκηση και το Κοινοβούλιο στο Λουξεμβούργο. Αντιπροσωπείες από την Επιτροπή μας επίσης επισκέφτηκαν, ε, ε, ε, άλλες χώρες. Είχαμε επίσης στη ληστούς ε, συναδέλφους σας υπουργού ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο απάντησαν όλοι εκτός από την Βουλγαρία, την Δανία και τη Σλοβενία. Το λέω δημοσίω γιατί θα ήθελα να το μεταφέρουν οι ευρωβουλευτές που προέρχονται από αυτές τις χώρες στις κυβερνήσεις τους έτσι ώστε να ε, λάβουμε τις απαντήσεις αυτών και τριών κυβερνήσεων όσο το δυνατόν συντομότερα. Θα ακούσουμε λοιπόν την παρουσίαση του Προέδρου του ΕΚΟΦΗΝ. Θα μας ενημερώσει που βρίσκεται η συζήτηση επί του κειμένου που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα tax rulings, για αυτές τις αποφάσεις φορολογικού χαρακτήρα. Μια ανακοινωσία που έγινε από την Επιτροπή τον ε, Ιούνιο και άλλες πρωτοβουλίες που έχουν πολύ μεγάλη σημασία, όπως η πρωτοβουλία BEPS στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ. Κατόπιν θα δώσω το λόγο στον εισηγητή και σε άλλα μέλη της Επιτροπής. Έχουν εγγραφεί στον κατάλογο 12 ομιλητές. Θα ζητήσω από ε, τους συναδέλφους να τηρήσουν τον χρόνο των δύο λεπτών για κάθε ομιλητή. Δυστυχώ πρέπει να είναι μικρό αυτό ο χρόνο, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των ανθρώπων που έχουν εγγραφεί στο κατάλογο και επίση γεγονότο ότι στι 6 ακριβώ θα πρέπει να ξεκινήσουμε τι ακροάσει των Υπουργών. Κύριε ε, Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, με χαρά χαίρομαι που είμαι παρόν σήμερα εδώ και θα σα δώσω μια εικόνα για το που βρισκόμαστε στα φορολογικά θέματα. Έχετε το σχέδιο έκθεσης για το επιθετικό προγραμματισμό, φορολογικό προγραμματισμό από επιχειρήσεις που είναι ψηλά στην ημερήσια διάταξη των κρατών μελών και της Ένωσης του ΩΣΑ και της ομάδας των 20. Το Λουξεμβούργο ως προεδρεύουσα χώρα της Ένωσης έθεσε την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην υψηλότερη θέση των προτεραιοτήτων της και είναι στη μέση διάταξη και των, του ΕΚΟΦΗΝ τους τελευταίους δύο μήνες όπως ξέρετε. Οι δραστηριότητες της Ένωσης στον τομέα αυτό επιταχύνθηκαν εν πολλής, διότι και οι Υπουργοί Οικονομικών συμφωνούν όλοι ότι δεν μπορούν να συμφωνεί, να, δεχθούν την απώλεια εσόδων, ιδίω σε περιόδους ε, δημοσιονομικών περιστολών, όταν οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν περισσότερους φόρους και ζητούν δίκαιη κατανομή της ε, φορολογικής επιβάρυνσης. Στην όλη συζήτηση για τα θέματα φορολόγησης υπάρχουν χώρες και πολίτες που τονίζουν το θέμα αφενός ε, του φορολογικού ανταγωνισμού και από την άλλη άτομα που ζητούν οι επιχειρήσεις να πληρώνουν το δίκαιο βάρος των φόρων. Οι δύο αρχές αυτές είναι αρχές πάνω στις οποίες πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Πώς αυτό γίνεται στο Συμβούλιο. Αφενός προσπαθώντας να επέρθει συμφωνία για ουσιαστικό δίκαιο με οδηγίε, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούμε και το soft law, όπως τον κώδικα δεντολογίας. Σε αυτή την πραγματιστική προσέγγιση, η Προεδρία ετοίμασε ένα νοδικό χάρτη συνολικό για τα BEPS ήδη τον Ιούλιο, ούτω ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στη δουλειά μας. Οι προβλεπόμενες δράσεις βράχη πρόθεσμα όλες έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται στους πρώτους, ε, κατά τους πρώτους μήνες της Προεδρίας. Αυτό αφορά και ειδικά νομοθετικά κείμενα, την οδηγία για την ε, αυτόματη ανταλλαγή αποφάσεων ή τον ε, ενιαίο φόρο επιχειρήσεων, την οδηγία για τα royalties, αλλά και για οριζόντια θέματα όπως το ελάχιστο αποτελεσματικό φορολογικό βάρος. Η εντολή που έχει δοθεί στην Φορολογική Επιτροπή υπογραμμίζει και τη δική σας δουλειά στο συγκεκριμένο θέμα για τα rulings και συναφή μέτρα. Οι φορολογικές αποφάσεις, τα tax rulings, είναι πολύ σημαντικά και για το Συμβούλιο. Η έγκριση της οδηγίας ε, που έχει τα, ε, τα το τίτλο DAC 3 είναι βασικός μας στόχος και θα επανέλθω στο θέμα αυτό αργότερα. Γνωρίζετε φαντάζομαι ότι δεν θα μπορέσω σήμερα να σας μιλήσω για το τι κάνει κάθε κράτος μέρος χωριστά για τις παρεμβάσεις, ούτε για θέματα κρατικών ενισχύσεων που επίσης καλύπτονται από την Επιτροπή, ιδίως την κυρία Φεστάγκερ, αλλά θα μπορούμε να συζητήσουμε για το τι κάναμε και θα κάνουμε στο Συμβούλιο μέχρι το έτος της Προεδρίας του Λουξεμβούργου, το τέλος της Προεδρίας του Λουξεμβούργου, συγγνώμη. Θα σταθώ λίγο περισσότερο λοιπόν στις δραστηριότητε του Συμβουλίου. Βλέπω στο κείμενο του σχεδίου σας ότι η Επιτροπή καλωσορίζει την έγκριση της οδηγίας μητρικών θηγατρικών και δίνεται ταυτόχρονα έμφαση στην οδηγία για τόκους και royalties που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί αλλά επί τις οποίες ε, δουλεύουμε με σκληρό τρόπο. Πέραν τη προσοχή που δίνουμε στην καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή και αποφυγή, το Συμβούλιο αποφασισμένο να δράσει και κατά των ε, αθέλητων συνεπειών της φοροαποφυγή ή της, του επιθετικού φορολογικού προγραμματισμού, δηλαδή την, ε, παρά, την αθέμητη χρήση νόμιμων τρόπων για να μην πληρώσει κάποιο φόρου ή να πληρώσει λιγότερου φόρου. Προ τούτο οι Υπουργοί στην ευκαιρία τη άτυπη συνάντηση του ΕΚΟΦΗΝ στο Λουξεμβούργο στις 11 Σεπτεμβρίου είχαν μια καρποφόρα συζήτηση για την ελάχιστη αποτελεσματική φορολόγηση, συζήτηση που θα χρησιμεύσει ως βάση για τη μελλοντική δουλειά. Θέλω να εξηγήσω πού βρισκόμαστε τώρα στο, στους πιο σημαντικούς φακέλους. Ξεκινώ με, τις με τη βασική προτεραιότητα. Την πρόταση οδηγίας για τις φορολογικές αποφάσεις, tax rulings. Η τεχνική ανάλυση της Επιτροπής ε, συνεχίζεται ακόμα. Το Συμβούλιο, ωστόσο, έχει πρόθεση να προχωρήσει γρήγορα για αυτές τις σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των, της άτυπης συνάντησης του ΕΚΟΦΗΝ στο Λουξεμβούργο και σύμφωνα και με τις συστάσεις της Επιτροπής σας, η Προεδρία θα προσπαθήσει να επιτύχει πολιτική συμφωνία για αυτόν τον σημαντικό φάκελο στο επόμενο ΕΚΟΦΗΝ στις 6 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει έγκριση της οδηγίας πριν το τέλος του 2015. Αυτός είναι ένας πολύ γρήγορος τρόπος να προχωρήσουμε λοιπόν όταν σκέφτεστε ότι η οδηγία αυτή υποβλήθηκε μόνο την Άνοιξη φέτος. Ενοποιημένη φορολογική βάση τώρα ε, των για τις τα κράτη-μέλη θέλουν να σταθούν ιδίω στις διεθνείς διαστάσεις anti-BEPS της πρότασης αυτής. Η Προεδρία άρχισε να συζητά τα θέματα αυτά που γίνονται όλο και σημαντικότερα μετά την πρωτοβουλία BEPS του ΟΣΑ που ο Σονούπο καρποφορεί. Όπως ανέφερε και η συγκήτρια στο σχέδιο έκθεσης, το, η δουλειά σχετικά με τα BEPS στην Ένωση και το αντίστοιχο έργο του ΩΣΑ είναι συμπληρωματικά ο συντονισμός που στο παρελθόν ήταν επιτυχής συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και η Προεδρία μας κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει. Σε ό,τι αφορά την οδηγία τόκι και royalties, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μετά την συζήτηση τον Ιούνιο, το... η Προεδρία υπέβαλε πρόσφατα νέες ε, προτάσεις προς συζήτηση στο τέλος του μήνα για να υπάρξει πρόοδος κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων. Για το οριζόντιο θέμα, οριζόντια ελάχιστη αποτελεσματική φορολόγηση. Η Προεδρία θέλει να γίνει συζήτηση για το οριζόντιο αυτό ζήτημα, ιδίω στο πλαίσιο τη οδηγία για τους στόκους και τα, και Εκεί θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτή η έννοια. Και για το λόγο αυτό βάλαμε στη μέση διάταξη του άτυπου εκοφήν πολύ τολμηρό εγχείρημα, γιατί ξέρουμε πόσο ευαίσθητο είναι το συγκεκριμένο ζήτημα. Πίστεψε ότι, ήταν μια καλή, ότι είχαμε μια καλή πρώτη συζήτηση για το θέμα, η οποία αποκάλυψε και πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα της ελάχιστης αποτελεσματικής φορολόγησης, θα εξετάσουμε ποιες δυνατότητες υπάρχουν στο εγγύς μέλλον να συμπεριλάβουμε την έννοια αυτή στην οδηγία των ε, τόκων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ομάδα τώρα για τον κώδικα διοντολογίας εξετάζει τώρα το standstill και το rollback των, των ε, ζημιογόνων ε, φορολογικών καθεστώτων τα κριτήρια τώρα, η ομάδα για τα κριτήρια έναντι των τρίτο χρόνο προχωρά και τώρα μπαίνουμε σε ένα πιο αποτελεσματικό διάλογο με το Λίχτενστάιν για τα θεωρούμενο ζημιογόνα καθεστώτα. Αυτή τη στιγμή ωστόσο πιστεύουμε ότι προχωράει η δουλειά και στο κώδικα διοντολογίας, κάτι που αντικατοπτρίζεται και για το μέλλον τη ομάδα αυτή. Ο στόχο είναι να μπορέσει να αντιμετωπίσει τι νέε προκλήσει που αφορούν το τομέα των ΠΕΠΣ με αποτελεσματικό τρόπο και θα εκμεταλλευτούμε την επιτυχημένη δουλειά που έκανε η ομάδα αυτή εδώ και πολλά χρόνια προσπαθώντα να δούμε πώ μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στο μέλλον. Ξέρω και το σημειώνω ότι οι εμπειρογνώμονε έχουν δουλέψει ε, αποτελεσματικά για την αναθεώρηση του προγράμματο εργασία του κώδικα. Τελευταίο θέμα που θέλω να αναφέρω αφορά στις τρίτες χώρες. Ζούμε σε, μια παγκοσμιοποιημένη εποχή, εποχή, οπότε στην ομάδα εργασία υψηλού επίπεδου για τις αρχές της καλής διακυβέρνησης στα φορολογικά θέματα έχουν γίνει συζητήσεις... για το πώς οι αρχές αυτές μπορούν να προωθηθούν και σε τρίτες χώρες. Πιστεύουμε ότι αυτό α, αξίζει να συζητηθεί περαιτέρω στο Συμβούλιο και στην ομάδα εργασία υψηλού επίπεδου, γιατί η Ένωση έχει ένα ευρύ φάσμα συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολόγησης και εφόσον η οικονομία παγκοσμιοποιείται. Ελπίζω ότι οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες και σας δίνουν καλή επισκόπηση της κατάστασης. Είμαι αποφασισμένο να συζητήσω τα θέματα φορολογίας του ΕΚΟΦΗΝ, προωθώντας τα περισσότερο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, με έναν συνολικό τρόπο, αναζητώντας τη σωστή προσέγγιση στην φορολογική πολιτική της Ένωσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν θέλουμε να δούμε την ε, αύξηση των εσόδων αφενός, αλλά τη δημιουργία ανάπτυξης θέσεων εργασίας και ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη στα πλαίσια μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Η φορολογία είναι στην καρδιά όλων αυτών των θεμάτων και με χαρά περιμένω να συζητήσουμε το θέμα αυτό μαζί. Euh, σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπω ε, σα ανέφερα ε, πρέπει να προσέξουμε τη διαχείριση του χρόνου γιατί είναι 5 και 20 και στι 6 θα ξεκινήσουμε ε, την ακρόαση των Υπουργών. Υπάρχουν 12 εγγεγραμμένοι από τους συζητητές και σκιώδεις συζητητές και δύο εκπρόσωποι των ε, πολιτικών ομάδων. επιδομένως θα ήθελα να συζητήσω ζητήσω δύο λεπτά ο καθένας να μιλείτε. Για να δώσουμε την ε, δυνατότητα και στον πρόεδρο Γκράμενια να απαντήσει. Πριν δώσω την, το λόγο στον εισηγητή, μιας και αναφερθήκατε στις εργασίες ε, της ομάδας εργασίας για την κώδικα διοντολογίας. Εμείς επιθυμήσαμε να, να δεχτούμε να λάβουμε την έκθεση των πρακτικών αυτής της ομάδας εργασίας. Γνωρίζουμε τους θεσμικούς προεπεριορισμούς, μιας και πρόκειται για μια διακυβερνητική ε, ομάδα εργασίας κτλ. Και δυστυχώς δεν έγινε δεκτό το αίτημά μας. Απευθυνθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει στην κατοχή της αυτά τα έγγραφα αν και η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι τα έγγραφα αυτά είναι στην ιδιοκτησία των κρατών μελών, ανήκουν στα κράτη-μέλη, επομένως η Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα να μας τα αποστείλει. Θα ήθελα να σας ζητήσω λοιπόν να ασκήσετε πιέσεις εσείς ε, με τις προσβάσεις που έχετε στο Συμβούλιο Υπουργών και πιθανώς και στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου έτσι ώστε να λάβουμε αυτές τις πληροφορίες. Δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο στην Ελίζα Φερέιρα, μία από τους δύο συγητές μας που σίγουρα την γνωρίζετε, γνωρίζετε επειδή σας επισκέφθηκε στο Λουξεμβούργο. Ελίζα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε ε, Υπουργέ, θα σας θέσω το ερώτημά μου στα αγγλικά γιατί αισθάνομαι πιο άνετα στη γλώσσα αυτή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα ήθελα να καταλάβω καλύτερα πώς έχουν εξελιχθεί οι συζητήσεις μέχρι τώρα και κατά πόσον υπάρχει πιθανότητα ε, να ε, αλλάξει η αντιμετώπιση των ζητημάτων φορολογικών αποφάσεων τύπου tax ruling, μια και ξεκίνησαν αυτέ οι πρωτοβουλίε από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά την ανισότητα που υπάρχει ανάμεσα στη φορολογική βάση, οι άμεσε ξένε επενδύσει στο Λουξεμβούργο ανέρχονται στο 424% του ΑΕΠ και 5.206% του ΑΕΠ. Επομένως, αυτές οι ανισορροπίες που είναι προφανείς από το παρελθόν έχουν συζητηθεί στο Συμβούλιο γιατί έχετε συζητήσει πώς αυτές τις καταστάσεις θα τις αποφύγουμε στο μέλλον. Επίση, υπάρχει η πιθανότητα να βρεθεί μια συμφωνία στο ζήτημα του πακέτου για τη διαφάνεια και αν ναι, θα ήθελα να ξέρω περισσότερε λεπτομέρειε. Γιατί ένα, μια συμβαστική λύση, μια συμφωνία μπορεί να είναι καλή ή όχι. Επίσης, ποια θα είναι η περίοδος αναδρομικής ισχύως που προβλέπετε ε, για την ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών. Επίσης, ποιε θα είναι οι αρχές που θα το υλοποιήσουν αυτό και πότε προβλέπεται η ημερομηνία θέση στην εφαρμογή αυτής της νέας συμφωνίας. Τι ακούγεται στο Συμβούλιο, δεδομένου ότι πλησιάζουμε στην 6η του Οκτωβρίου. Τελευταίο σχόλιο. Τι πιστεύετε για τους φορολογικούς παραδείσους. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να έχουμε κάποια ευρωπαϊκά κριτήρια, τα οποία να πηγαίνουν ίσω και ένα βήμα παραπέρα από τα κριτήρια του ΟΑΣΕ για του φορολογικού παραδείσου, όπω για παράδειγμα εκείνα που προτείνουμε στην εκθεσή μα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Λίζα και σα ευχαριστώ επίση που ε, κρατήσατε και το χρόνο. Δίνω το λόγο στον κύριο Μίκαελ Τόιρερ, τον άλλο συνεισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Καμάνια, ως ε, εκπρόσωπε της ε, Προεδρία Λουξεμβρού. Είναι πολύ σημαντικό που ήρθατε εδώ και είναι εξάλλου και μία, ένα μήνυμα ότι μας παίρνετε στα σοβαρά. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα ήθελα να αναφερθώ στα έγγραφα. Ως Κοινοβούλιο ζητήσαμε έγγραφα μεταξύ άλλων τα πρωτόκολλα που ζήτησε ο Πρόεδρος, ε, τον κώδικα συμπεριφοράς, οι ιδεοντολογίε, αλλά και άλλα έγγραφα που αναφέρεται η θέση της Επιτροπής. Αυτά τα έγγραφα μας λέτε δεν μπορείτε να μας τα δώσετε γιατί δεν συμφωνεί το Συμβούλιο και εμποδίζει κάτι τέτοιο. Εγώ το θεωρώ απαράδεκτο ότι δεν μπορούμε να δούμε, ούτε καν να δούμε αυτά τα έγγραφα, προφανώ και τηρώντας ε, την αρχή της ε, χεμίτιας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόσο στην Επιτροπή Ελέγχου Προπλογισμών έχει δει έγγραφα της ε, Όλαφ, όσο και στην ΕΚΟΝ μπορέσαμε να δούμε μυστικά έγγραφα της ΕΚΤ. Γιατί λοιπόν δεν μπορείτε να μας τα δώσετε να τα δούμε. Νομίζω ότι αυτά σημαίνει ότι δεν δέχεστε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και αυτό είναι Το δεύτερο που θέλω να θίξω αφορά στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Με βάση λοιπόν τις πληροφορίες που έχω εγώ, Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά κρατών μελών που αντιτίθενται στην νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσπαθούν, αν θέλετε, να βελτιώσουν ουσιαστικά αυτή την πρόταση. Υπάρχει λοιπόν και η τοποθέτηση του Bundesrat, της Δεύτερης Βουλής της Γερμανίας, που δεν δέχεται η Κομισιόν να διατηρεί τα text rulings. Η πρόταση της Γερμανίας είναι ε, να δίδονται αυτά τα έγγραφα ανώνυμα εδώ όμω θέλω να πω ότι υπάρχει αντίδραση από την Ισπανία. Με βάση τις πληροφορίες που έχω, η Ισπανία επιθυμεί να δίδονται μόνο στατιστικές πληροφορίε για τα text rulings και από ό,τι φαίνεται η Μεγάλη Βρετανία είναι επιφυλακτική έτσι κι αλλιώ. Ερωτώ λοιπόν, ισχύουν αυτά που λέω και πώς θα μπορέσουμε η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών να προχωρήσει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η Κομισιόν να έχει πραγματικά τη δυνατότητα της, ε, του ελέγχου. Εσείς επίσης επισημάνατε τον ΟΣΑ. Δεν θέλουμε όμως να έχουμε ε, αδέσμευτες συστάσεις, να έχουν συστάσεις νομοθετική ισχύ. Αναφέρεται ότι Υπάρχει ε, μία συμφωνία της ε, Γερμανίας ε, σχετικά με τον ΟΣΑ, του Λουξεμβούργου όμως μόνο περιορισμένη συμφωνία. Τι έχετε να πείτε από αυτού. Ευχαριστώ πολύ τους συζητητές. Ο κύριος Γιούναρ Χόκμαρκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτό που είναι απόλυτα σαφές είναι ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την φόρο αποφυγή και επίσης να αποφύγουμε την ε, φοροαποφυγή η οποία κατά κύριο λόγο στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Υπάρχουν και άλλοι πολύ επιζήμιοι τρόποι που μπορεί να προκύψουν μέσα από την νομοθεσία. Πάντως είναι και σημαντικό γενικά να έχει κανείς μια εικόνα. Το λέω αυτό διότι μερικές φορές τα κράτη-μέλη τίνουν με χαμηλότερο εταιρικό φόρο ή άλλες με υψηλότερο εταιρικό κάτω από το αναπτυξιακό πρίσμα να δίστανται, αλλά αυτό δεν είναι σημαντικό και δεν είναι αλήθεια, γιατί όλοι θέλουν να έχουν περισσότερες επενδύσεις. Και είναι αλήθεια ότι Όσο υψηλότερος είναι ο εταιρικός φόρος στα κράτη-μέλη, τόσο περισσότερο τα κράτη-μέλη προσφέρουν εκπτώσεις και παρατηράκια στον νόμο, όπως λέγονται. Ας δούμε λίγο τα διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν αυτά που έχουν, ας πούμε, ε, ένα εφάπαξε συντελεστή, χαμηλότερους ε, ε, χαμηλότερη φορολογία. Αυτοί όμως έχουν περισσότερα έσοδα από άλλα που έχουν υψηλότερου συντελιστέ που όμως σας είπα χορηγούν εκπτώσεις και παραθυράκια. Εσείς τώρα πώς θα διαμορφώσετε τη συζήτηση ε, που δεν πρέπει να οδηγήσει ε, σε υψηλό φόρο γιατί αυτό όπως σας είπα πολλές φορές οδηγεί στη φοροαποφυγή. Μας ενδιαφέρουμε να έχουμε χαμηλούς εταιρικούς φόρους που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης που έτσι και αλλιώς σας είπα αποτελούν εγγύηση για την εισπραξιμότητα των φόρων. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να τοποθετήσετε τη συζήτηση σε σωστό πλαίσιο. Ακριβώς δύο λεπτά μίλησα, Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστώ, Γιουνάρ. Για την ομάδα S&D, η κυρία Καϊλή. Δύο λεπτά. Thank you. Excuse my voice, but we had elections in uh, Greece. Ευχαριστώ, ζητώ συγγνώμη για την φωνή μου. Φταίνει οι εκλογές στην Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε του Κοφίν. Έχω την Εξή ερώτηση. Στι 17 Ιουνίου ανακοίνωσε η Επιτροπή ένα νέο σχέδιο για μια πιο δίκαιη φορολόγηση των επιχειρήσεων στην ε, Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι στο Λεξεμβούργο η οικονομία έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην προσέλκυση επενδύσεων εξαιτία του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτου, το οποίο οδηγεί σε μια χαμηλή φορολόγηση εισόδων τα οποία θα έπρεπε να είχαν ε, τύχη φορολόγηση σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Θα ήθελα να σας, να σας ρωτήσω λοιπόν τι έχετε κάνει για να προωθήσετε τη διαφάνεια ε, και τη διαφανή συζήτηση ε, επί αυτού του σχεδίου δράσης της Επιτροπής και επίσης γιατί δεν έγινε δημόσια συζήτηση στο Συμβούλιο πάνω σε αυτό το σχέδιο για την αποτελεσματική φορολόγηση, έτσι ώστε να ακούσουν και οι πολίτε τη Ευρώπη ποια είναι η θέση κάθε κράτου μέλου, ποια είναι η θέση του Υπουργού τη χώρα του, γιατί αυτή η συζήτηση έγινε ε, πίσω από κλειστέ πόρτε του ΕΚΟΦΗΝ. Επίση, και η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επισημάνει τη σημασία τη διαφάνεια όσον αφορά την φορολόγηση των επιχειρήσεων και ακόμα περισσότερο των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν ζήτησε να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία που να συζητηθεί ε, στο πλαίσιο της ε, οδηγίας ε, για τους μετόχους στο Συμβούλιο να ζητηθεί από τις εταιρείες να δημοσιεύουν τους μετόχους τους και τα μυρίσματα που λαμβάνουν αυτοί σε κάθε μια από τις χώρες τις οποίες λειτουργούν, δραστηριοποιούνται αυτές οι εταιρείες. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι ποιες είναι οι συγκεκριμένες ενέργειες που προβλέπει η Προεδρία του Λουξεμβούργου, έτσι ώστε αυτές οι υποχρεώσεις να συμπεριληφθούν για τις εταιρείε στην ε, οδηγία τη σχετική. Να είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε και να φροντίσουμε να καταπολεμήσουμε την επιθετικό φορολογικό ε, προγραμματισμό από αυτές τις εταιρείε. Για το ECR, ο κύριος Κράσνοντεψκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις. Αλλά στα πολωνικά καλύτερα, για μένα. Σας δίνει πολύ ωραία γλώσσα τα πολωνικά. Φορέστε ακουστικά λοιπόν. Έχουν ωραίο ήχο και καλό είναι να θυμό θυμόμαστε τον ήχο αυτό που και που. Ένα σχόλιο καταρχάς. Αυτό που συχνά ξεχνάμε στις διαπραγματεύσεις είναι ότι η φορολογική πολιτική είναι βασικό στοιχείο των οικονομικών, των εθνικών οικονομικών πολιτικών. Για να υπάρχει λοιπόν θεμητός ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων από χώρα σε χώρα θα πρέπει να υπάρχει θεμητό δίκαιο φορολογικό σύστημα σε όλη την Ευρώπη. Η ερώτηση που θέτουν είναι εξής. Το ECOFIN υιοθέτησε μια σειρά κανόνων για την ε, φορολογία επιτρέποντας ταυτόχρονα και στις εθνικές κυβερνήσεις να έχουν ανταγωνιστικές οικονομίες και φορολογική πολιτική. Μπορεί να γίνει αυτό. Δεύτερον, όσα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων η Επιτροπή έθεσε ως πανάκια την, το, τον τρόπο με τον οποίο ο φορολογικός προγραμματισμός θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τη φοροαποφυγή. Αυτό κατά την άποψη πολλών εμπειρογνωμόνων, είναι λάθος. Πώς, ε, από πού αντλείται εμπειρογνωμοσύνη για τις προτάσεις που κάνετε για να πετύχετε τους στόχους που έχετε θέσει. Πώς λαμβάνετε υπόψη τις διαφορές των κρατών μελών στο ΕΚΟΦΗΝ. Ευχαριστώ. Για τους φιλελεύθερους, ένα λεπτό, ο Μιχαήλ. Κύριος ε, Τόιο, ε, κοιτάξτε, δεν μπόρεσε να έρθει αδελφός μου, γι' αυτό λοιπόν την αντικαθιστώ και ένα πολύ σύντομο ερώτημα. Κύριε Υπουργέ, δείξατε το θέμα της ε, ελάχιστης φορολογίας, ελάχιστο tax rate, όπως λέγεται, το συμπεριλάβαμε αυτό στην εκθεσή μας και μετά από πολλές συζητήσεις με την συνάδελφο κυρία Φερέρα, αυτή ήταν η δική μου η για να συνενέσω να συμπεριλαμβάνεται και μέγιστο tax rate, maximum tax rate. Η ΟΣΑ προβλέπει και αυτός ένα μέγιστο τέτοιο φορολογικό συντελεστή. Βεβαίως ε, το να υπάρχουν ε, αρνητικά κίνητρα για την ε, φοροαποφυγή, αποφυγή, αυτό είναι σημαντικό εμείς καταθέσαμε μια ισορροπημένη πρόταση. Η πρόταση ήδη συζητήθηκε από το Συμβούλιο και ερωτώ εσείς όσον αφορά τα μέτρα τα φορολογικά, της φορολογικής απλούστευσης του ΩΣΑ, ποια είναι η δική σας συγγνώμη. Äh, Όταν ήμασταν, λέει ο κ. Φάμπιο Ντεμάζη, σε εσά και σας επισκεφθήκαμε, ε, ακούσαμε ότι ε, οι φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου έχουν απευθυνθεί στη Γερμανία και στη Γαλλία ε, για πολύ ψηλά κέρδη τα οποία ε, αναφέρονται στο Λουξεμβούργο και ρωτώ κατά πόσον χωρίς να μπείτε σε μεμονωμένες περιπτώσεις, μπορείτε να μας πείτε τις προειδοποιήσεις που κάνατε προς τη Γαλλία και τη Γερμανία, τον αριθμό των προειδοποιήσεων για πολύ ψηλά κέρδη, αυτό θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για να μην εστιάζει τη συζήτηση μόνο στο Λουξεμβούργο. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι γιατί ε, το Λουξεμβούργο από το 2015 έχει υπογράψει οκτώ συμφωνίες διπλής φορολόγησης μεταξύ άλλων με, τα, με τις νήσους Μαν, με τη Σιγκαπούρη και πολλούς άλλους. Ε, ποια είναι λοιπόν η δική σας η προτεραιότητα όσον αφορά αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους. Και τέλος θα ήθελα να γνωρίζω το εξής. Στις 14 Σεπτεμβρίου υπήρξε μία συζήτηση για τα δικαιώματα των μετόχων και τις ε, καταχώρες συστάσεις. Εσείς ε, λοιπόν παρακαλέσατε τα κράτη-μέλη να τοποθετηθούν στο πλαίσιο αυτής της ε, αναχώρα συστάσεις με non-paper. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι η θέση της Επιτροπής αλλά και της δικής σας της κυβέρνησης ο κύριος Μοσκοβισή είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι αυτές οι χώρα συστάσεις καλό είναι να δημοσιοποιηθούν, αλλά διαφωνεί η Κομισιόν. Και γι' αυτό με ενδιαφέρει. Εσείς μίλησατε με τον κύριο Γιούγκερ για το θέμα αυτό. Συμφωνεί ε, με αυτή την, αντίδραση. Τι λέει. Η μόλις για τους πράσινους. Κύριε Υπουργέ, τα στοιχεία δείχνουν ότι από τότε που έγινε υπουργό οικονομικών ε, τη χώρα, ο κ. Γιούνκιο το 1981, δεν ανέβηκε η φορολογία από το 0% στο 10%. Η χώρα σα εξαρτάται κατά συνέπεια στο έντονα στο σύστημα φοροαποφυγής μεταφοράς κερδών. Η οικονομία σας εξαρτάται από τις δραστηριότητε αυτές που κατά την άποψή μου τουλάχιστον δεν έχουν κοινωνικά ε, πλονεκτήματα. Ποια στρατηγική έχετε για να περάσετε από μια εποχή φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ κρατών σε μια υγιή νομοθετική φορολογική πολιτική. Ο Αντιάντελ Τελτούρ ε, που παρουσίασε, που δημοσιοποίησε μια σειρά ε, στοιχείων των, του για τις φορολογίες του Λουξεμβούργου δικάζεται αυτή τη στιγμή. Αν δεν μας είχε προειδοποιήσει γι' αυτά, δεν θα ξέρουμε τίποτα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τη Επιτροπή, η Επιτροπή μας διαπίστωσε ότι το νομικό πλαίσιο προστασία ε, από τη φοροαποφυγή του Λουξεμβούργου δεν είναι επαρκής. Είναι σωστό να δικάζεται κάποιο ο οποίος απελευθέρωσε πληροφορίε προς το όφελος του κοινού καλού. Μια τελευταία ερώτηση προ εσά ω προεδρεύοντο τη Ένωση είπα, ζητήσατε, είπατε μάλλον στην Επιτροπή ότι είστε υπέρ τη μεγαλύτερη διαφάνεια στα φορολογικά ζητήματα. Θα ξεκινήσει ένα τρίλογο για, για την οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων. Όπου εμεί υποστηρίζουμε την ε, ε, αρχή τη αναχώρα δημοσιοποίηση ε, και λογοδοσία. Θα υποστηρίξετε την δημόσια ανακοίνωση χώρα με χώρα των φορολογικών κερδών στις διαπραγματεύσεις ή θα οδηγήσετε εκ νέου σε καθυστέρηση αυτών των ε, δυνατοτήτων που περιμένουν και προσδοκούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ευχαριστώ συνάδελφε. Για το EFDD, ο κύριο Σέμπτη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να ασχοληθώ με κάποια θέματα που δεν ε, εφήγησαν ακόμα από τους συναδέλφους. Πρώτον, ο ρόλος των τραπεζών. Γνωρίζουμε ότι στις ε, δίκες για την φοροποφυγή και φοροδιαφυγή είναι καθοριστικός ο ρόλος των τραπεζών και εντός και εκτός Ένωσης και ως σύμβουλοι των πολυεθνικών και ως διαχειριστές ε, και υπεύθυνοι των συναλλαγών διότι όλες οι ροές ε, χρημάτων νομίμων και μη περνούν μέσω τραπεζών. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το Συμβούλιο πέραν των συζητήσεων για συστάσεις που προέκυψαν από την ομάδα εργασίας για τα BEPS συζητά και το ενδεχόμενο μεγαλύτερου ελέγχου και διαφάνειας των τραπεζών ακριβώς ε, σε αυτή τη δραστηριότητα. Κάτι άλλο που θέλω να ξέρω είναι συζητείται στο Συμβούλιο το θέμα των σχέσεων μεταξύ κρατών μελών και άλλων εδαφών ε, ελεγχόμενων από ένα κράτος ή παλιών απικιών. Από ό,τι προέκυψε σε ακροάσεις που κάναμε εδώ, ανέκυψε ε, σαφείς σαφής σχέσεις μεταξύ του ρόλου που παίζουν διμερείς συμφωνίες ε, μεταξύ κρατών μελών της Ένωσης και παλαιών εδαφών τους που επιτρέπουν στο μεν κράτος μέλος τυπικά να σέβεται την νομοθεσία, αλλά να την καταστρατηγεί με αυτές τις διμερείς ε, συμφωνίες. Ε, υπάρχει συζήτηση για μια ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ αυτών των κρατών και των ε, λοιπόν ε, εξαρτημένων εδαφών. Τώρα, το aggressive tax ruling, ο ορισμός αυτός, είναι διαφορετικός από χώρα σε χώρα. Μήπως δουλεύετε σε επίπεδο συμβουλίου για να καταλάβετε πραγματικά τι σημαίνει aggressive tax ruling. Ποιο είναι το επίπεδο που χρειάζεται. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει για να τύχει ομοιόμορφο ορισμό. Ευχαριστώ Μάρκο. Η κυρία Μπάρμπαρα Κάπελ για το ΕΝΕΦ. E Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ και Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Στην αρχική σας παρέμβαση ε, μας παρουσιάσατε ορισμένα σημαντικά θέματα τα οποία ε, συζητούνται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο κατά προτεραιότητα. Δηλαδή το CCTB, η οδηγία περί ε, αδειοδοτήσεων και παρεμφερή. είπατε ότι την επόμενη φορά, τον Οκτώβρη, το Συμβούλιο θα συνεδριάσει στο Λουξεμβούργο και γι' αυτό θέλω να σας παρακαλέσω μερικά πράγματα. Το Κοινοβούλιο έχει τρεις εκθέσεις που επεξεργάζεται και συνδέονται με αυτά τα θέματα που αναφέρατε. Έκθεση Φέρμπερ για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από την Επιτροπή ΕΚΟΝ και εδώ, κατά την άποψή μου, η σκιώδη εισηγήτρια έχει φίξει τρία βασικά θέματα που διαφοροποιούνται από αυτά που λέτε και εσείς και η Επιτροπή. Σύμφωνα λοιπόν με, την, με τον εισηγητή ε, δεν θα πρέπει ε, να ε, ελέγχονται μόνο τα διασυνοριακά συνοριακά ε, φορολογικά αδικήματα αλλά ε, και η σχετική ενημέρωση αλλά και όλα τα άλλα Επίσης, αυτό που αναφέρθηκε είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υπάρχει ένα κεντρικό αρχείο για όλες αυτές ε, τις ε, φορολογικές παραβάσεις και θέλω να ρωτήσω ποια είναι η άποψη του Συμβουλίου. Τώρα, το CCTB υπάρχει έκθεση Νίντε Μάια από το ECOFIN. Εκεί γίνεται λόγος ε, για, την επιθετική, για τον επιθετικό σχεδιασμό, φορολογικό σχεδιασμό, κυρίως όσον αφορά τις πολυεθνικές. Ξέρετε, αυτό το έχουμε πληροφορηθεί από, τα, από τις διάφορες διαδικασίες διαρροές. Θέλω λοιπόν από το εξή. Ε, μπορεί να υπάρχει για κάποιο χρονικό διάστημα το αφορολόγητο και να ξεφεύγει κανείς. Αυτό το συζητάτε ή όχι. Η τρίτη έκθεση είναι η έκθεση Φερέρα, το ΙΡΑΡ, η οποία συζητήθηκε και αναφέρθηκε εδώ. Ε, να υπάρχει λοιπόν ένα κεντρικό αρχείο, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, για text rulings και θέλω να ρωτήσω ποια ακριβώ είναι η στάση σας από αυτού. Ευχαριστούμε Μπάρμπαρα. το, για το ΕΛΚ ο κύριος Κίρτσος. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Προεδρία του Λουξεμβούργου κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, ωστόσο δεν είμαι σίγουρος ότι θα σας ακολουθήσουν όλες οι κυβερνήσεις. Και το ερώτημα είναι, θα υπάρξει μια πολιτική συμφωνία που χρειάζεται για αναθεώρηση των φορολογικού συστήματο ή μήπω θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου ορισμένε κυβερνήσει θα το αρνηθούν και αυτό θα υπονομεύσει την κοινή προσπάθεια. Επίση, θα ήθελα να ε, μου εξηγήσετε πιο αναλυτικά τη θέση σα για τα ζητήματα τη φορολογική κατοικία. Έχω την αίσθηση ότι πηγαίνουμε ε, προ ένα καθεστώ όλο και πιο ε, αυστηρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα δώσει θα βάλει σε πειρασμό τις πολυεθνικές εταιρείες να, να βάλουν την έδρα τους σε κάποιο κράτο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μπορούμε να το καταπολεμήσουμε αυτό γιατί διαφορετικά θα βρεθούμε σε μια κατάσταση που θα μειώσουμε τα φορολογικά έσοδα αντί να καταφέρουμε να τα αυξήσουμε. Ευχαριστούμε και τέλος κύριο Πορτάν για του Σοσιαλδημοκρατέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ευχαριστήσω τον Υπουργό του Λουξεμβούργου που ε, παρευρέθηκε στην συνάντησή μας και μας ενημέρωσε για την κατάσταση των συζητήσεων. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάει την φοροαποφυγή. Ταυτόχρονα ο ΑΣΕ έχει το πρωτοβουλία BEPS και ταυτόχρονα η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο διαδέχθηκαν στην Προεδρία την κυριόμενη του Συμβουλίου οι οποίες δύο αυτές χώρες, ε, κατά την άποψή μου, η Ορλανδία μάλλον, η Ορλανδία και η, το Λουξεμβούργο, έχουν μια ιδιαίτερη θέση, στο θέσω έτσι, στον τομέα της φοροαποφυγής. Εάν δείτε τις ξένες, άμεσες ξένες επενδύσεις, θα δείτε ότι το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία μαζί έχουν μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις από ότι το Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτό κάτι μας λέει. Έχω λοιπόν δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Συμφωνείτε για αυτήν την ιδιαίτερη θέση που έχουν λάβει η α, Ολλανδία και το Λουξεμβούργο στη διευκόλυνση της φοροαπολυφυγής. Ναι ή όχι. Και εάν ναι, συμφωνείτε μαζί μου ότι έχουν και ιδιαίτερη ευθύνη να την καταπολεμήσουν τη φοροαποφυγή αφού την διευκόλυναν. Δεύτερο ερώτημα. Δεν αναφερθήκατε στις εκθέσεις αναχώρα. Και γνωρίζουμε ότι αυτό έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο και ότι πολλά κράτη-μέλη, κάποια κράτη-μέλη μάλλον, έχουν αντιταχθεί στεναρά στη δημοσιοποίηση αυτών των εκθέσεων. Υπάρχει ακόμα αυτή η αντίσταση από την πλευρά του Συμβουλίου. Και αν ναι, ποια είναι η άποψή σα, πότε θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο για την οδηγία για του μετόχου Shareholder Directive και για τι συστάσει χώρα. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο για να απαντήσετε στα ερωτήματα των μελών τη Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πολλέ ερωτήσει. Θα προσπαθήσω να τις ομαδοποιήσω και ζητώ συγγνώμη αν δεν καταφέρω να τι αντιμετωπίσω όλε. ξεκινώ με αυτές που κανονικά δεν θα έπρεπε να απαντήσω, διότι εδώ είμαι πρόεδρος, ε, ε, ασκών την προεδρία του, του Ευρωπαϊκού του Συμβουλίου των Υπουργών. Πολλές ερωτήσεις αφορούσαν το Λουξεμβούργο. Να σας πω και εγώ δύο λόγια για το Λουξεμβούργο. Πρώτον, είχα δεχθεί την Επιτροπή Τάξης του Λουξεμβούργου και απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις που μου τέθηκαν. Εν πολλής, αυτό ικανοποίησε τις περισσότερες ε, από εσά. Συνεργαστήκαμε αρκετά και στείλαμε αρκετέ πληροφορίες στην Επιτροπή σας. Δεύτερο θέμα, διότι το ανέφερε ο προηγούμενος ομιλητής, ο κ. Στάν, για την χώρα και για μένα και τη δική μου. Υπογραμμίζω ότι το Λουξεμβούργο τους τελευταίους 20 μήνες άλλαξε ριζικά. Μεταρρυθμίσαμε πολλά πράγματα. Αλλάξαμε την νομοθεσία για την ανταλλαγή πληροφοριών μετά από αίτημα όπου δεν συμμορφωνόμασταν μέχρι τώρα και είμαστε αισιοδόξοι ότι θα συμμορφωθούμε σύντομα εμπολής. Αλλάξαμε το θέμα του τραπεζικού απορρίτου. Να υπογραμμίσω ότι, το ότι θεωρώ πολύ σημαντικό το θέμα της ε, ε, φορολογική μεταρρύθμισης. Ε, είναι στην πρόθεσή μας να συνεργαστούμε ουσιαστικά στο θέμα αυτό και νομίζω ότι κάνουμε μεγάλη πρόοδο στο θέμα αυτό. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά για τα θέματα της φορολόγησης και εδώ δεν μιλώ εξ ονόματος του Λουξεμβούργου αλλά εξ ονόματος της Προεδρίας αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι αρχές και η κυβέρνησή μου με έντιμο τρόπο προσπαθούν να συνεργαστούν μαζί σας. Για τα ερωτήματα που μου τέθηκαν με την ιδιότητα μου ως πρόεδρου. Το πιο επίγον, αυτόματη ανταλλαγή, ε, οδηγία για την αυτόματη ανταλλαγή αποφάσεων, tax rulings. Κανα δύο θέματα τέθηκαν πολλές φορές και οι συζητήσεις συνεχίζονται. Να σας πω λοιπόν ότι αισιοδοξώ πως σύντομα θα υπάρξει συμφωνία για την οδηγία αυτή. Κάνουμε ό,τι μπορούμε σε επίπεδο ομάδα εργασίας και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Πώς έλεγε ο Ντράγκη, whatever it takes, ώστε στις 6 Οκτωβρίου να κλείσουν τα θέματα που είναι κρεμή. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε για τι τις κάθε χώρα, αλλά νομίζω ότι όλες οι χώρε έχουν δεσμευθεί να υπάρξει συνένεση. Για το θέμα της αναδρομικότητας, η Επιτροπή είχε προτείνει να είναι αναδρομικό για 10 χρόνια, υπάρχει μια συνένεση για μια πενταετία. Όσον αφορά τον ρόλο της Επιτροπής, προχωρούμε προς μια κατεύθυνση όπου η Επιτροπή θα μπορεί να λάβει πολλές αλλά όχι όλες τις πληροφορίε. Καταλαβαίνετε προς τα που πηγαίνουμε. Αναγνωρίζετε ότι η Επιτροπή έχει ρόλο, όμως σε πολλές χώρες υπάρχουν κανόνες που εμποδίζουν να δίδονται όλες οι πληροφορίε στην Επιτροπή, ιδίως ονόματα. Αν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύο θέματα, θα προχωρήσει πολύ γρήγορα η οδηγία, που θα εφαρμοστεί επίσης πολύ γρήγορα. Και η ταχύτητα με την οποία εγκρίνεται η οδηγία αυτή, είναι επίτευγμα αυτό καθ' αυτό. Υπήρχαν ερωτήσεις για το πόσο βαθιά θέλουμε να μπούμε στις συζητήσεις για το τι σημαίνει aggressive tax ruling. Η οδηγία αυτή έχει σαν στόχο την αυτόματη ανταλλαγή. Σε συνέπεια τούτου θα γίνουν συζητήσεις για το τι σημαίνει αυτό το aggressive tax ruling βάσει της εμπειρίας που θα αντλήσουμε. Και η ομάδα του κώδικα δεντολογίας θα εξετάσει το θέμα αυτό. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που τέθηκαν σε ό,τι αφορά την αυτόματη αντιλογή αποφάσεων σε κάποια άλλα θέματα τώρα που είδα. Πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θεωρούμε όντως ένα πολύ σοβαρό εγχείρημα. Η κυρία Καηλή το ανέφερε. Και εξέφρασε και την λύπη της, διότι δεν ήταν δημόσια σχετική συζήτηση. Κάποιο άλλο το είπε. Α, και κάποιο άλλο μίλησε για το επί, ελάχιστο επίπεδο φορολογική επιβάρυνση. Πρέπει να σας πω ότι απετέλεσε, ε, ότι ήδη το ότι είχαμε αυτή τη συζήτηση ήταν ένα μεγάλο σημαντικό πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα ήταν μια άτυπη συνάντηση, διότι έτσι μπορέσαμε να το βάλουμε στην μερισσία διάταξη. Το θέμα έχει τεθεί, δεν μπορεί να μπει κάτω από το τραπέζι και θα επανέλθει στο θέμα των τόκων και δικαιωμάτων, των royalties. Αντί λοιπόν να λέμε ότι «Α, δεν τα κάνατε όλα». Δείτε το ανάποδα. Δείτε το ότι ήταν ένα θαραλέο πρώτο βήμα για να ξεκινήσει η σχετική συζήτηση. Σε πολλές χώρες, πολλές χώρες δεν σας πω, δεν ήταν ευτυχής που τέθηκε προς συζήτηση το θέμα αυτό. Η αναχώρα εκθέσεις. Και τι κάνουμε σχετικά. περιμένουμε τα αποτελέσματα της μελέτης αντικτύπου της Επιτροπής. Σε αυτή τη βάση θα δούμε πώς προχωράμε. Στο πλαίσιο αυτό τέθηκαν πολλές θεμητές ερωτήσεις, αλλά πρέπει να περιμένουμε την αξιολόγηση της Επιτροπής και πιθανές συστάσεις της. Το ερώτημα του Προέδρου για την πρόσβαση στα κείμενα, ιδίω ε, τη ομάδα κώδικα διοντολογία. Πρέπει να σα πω ότι καταρχήν το Συμβούλιο υποστήριξε τη διαφάνεια, αποστέλλοντά σα πολλέ πληροφορίε μέσω τη φορολογική ομάδα τη ομάδα φορολογία τον Μάιο. Και μάλιστα κάποια κράτη-μέλη και το Συμβούλιο εξέφρασαν επιφυλάξεις για την χορήγηση πλήρους πρόσβασης, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να υπονόμευε την υφιστάμενη πολιτική των κρατών και την καλή λειτουργία των ομάδων εργασίας. Αυτές είναι οι αρχές που δημιουργούν προβλήματα. Ο ρόλος μας ως προεδρίας είναι να βοηθήσουμε στην επίλυση του θέματος, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας θα συζητήσουμε για να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε μια ικανοποιητική λύση. Τι άλλο. Σχέσεις τρίτων χωρών, σχέσεις με τρίτες χώρες. και θέματα πώς φορούσαν στο ρόλο των τρίτων χωρών στην προτεσέλκιση εταιριών. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε στην Ευρώπη είναι να υπάρξει φορολογικός συντονισμός ή ένα φορολογικό σύστημα πιο κοντινό το ένα στο άλλο που θα προσαρμόζεται και στις πρωτοβουλίες BEPS. Γιατί το BEPS έχει πολλές ιδέες για, ε, για τον εξυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος στην Ευρώπη αφενός. Αφετέρου, αφετέρου εκτός Ένωσης, χώ, κάποιες χώρες εκτός Ένωσης πρέπει να τηρήσουν τους κανόνες των BEPS. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ένα στόχος ισότιμης, ισο, ισότιμη, ε, δίκαιης, ε, δίκαιο ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών η ερώτηση λοιπόν του τι θα γίνει στην Ένωση αν δεν υπάρξει κάτι τέτοιο, πρέπει να σας πω ότι η πρωτοβουλία BEPS ε δεν περιορίζεται στην Ένωση, είναι πρωτοβουλία της ομάδας των 20 και του ΩΣΑ για να υπάρχει μια πάνω κάτω ίση μεταχειρίση των επιχειρήσεων και να μην προσελκύονται επενδύσει για, φορολογικούς, για λόγους στην πραγματικότητα σε μια χώρα σε σχέση με μια άλλη. Μια τελευταία παρατήρηση. Περνάει και ο χρόνος. Τελειώνω λέγοντας ότι θα είμαστε σε επαφή μέχρι την ολοκλήρωση της έκθεσής σας. Αν έχετε και άλλες ερωτήσεις σε διμερές επίπεδο, να τις ε, συζητήσουμε και διμερός, διμερός. Όχι σήμερα, θα ήθελα να εκφράσω την επιθυμία να συνεργαστούν όλες οι χώρες με την Επιτροπή Τάξε και θέλω να τελειώσω με την παρατηρήση του Πρόεδρου εισαγωγικά. Κάποιες χώρες, λίγες, δεν έχουν στείλει καμία πληροφορία. Ε, ας ε, έχουμε μια ισότιμη αντιμετώπιση όλων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά διαβολική σύμπτωση, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που έχουμε ευκαιρία να προχωρήσουμε σε αυτά τα θέματα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Λουξεμβούργου. Δηλαδή να καταπολεμήσουμε κάποιες νομοθετικές πρακτικές οι οποίες είναι απαράδεκτες, αλλά ταυτόχρονα να καταλήξουμε σε ορισμούς ε, ενιών που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αξιοποιήσουμε την πρωτοβουλία BEPS από την πλευρά του ΑΣΕ. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε ε, η Προεδρία του Λουξεμβούργου να καταλήξει τον Οκτώβριο σε συμφωνία όσον αφορά την οδηγία για την ανταλλαγή πληροφοριών για να υπάρξει και τελική συμφωνία μέχρι το τέλος της χρονιάς σε άλλα θέματα όπως το CCCTB, καλό θα ήταν και εκεί να υπάρξει πρόεδρος. Αναφέρθηκε το ζήτημα από συναδέλφους και ευελπιστούμε να υπάρξει ε, συμφωνία από την πλευρά του ΕΚΟΦΗΝ πριν το τέλος της ε, Προεδρίας του Λουξεμβούργου και για το CCCTB. Τώρα, μιλώντας για την ανταλλαγή των αποφάσεων tax rulings και για την αναδρομική του ισχύ, ε, θα έλεγα ότι προσωπικά μιλάω τώρα είναι τελείως απαράδεκτο να παζαρεύουμε πόσο θα είναι η αναδρομική ισχύς. Ε, ε, θα... δεν είχε σημασία αν μιλάμε για μια απόφαση η οποία λήφθηκε πριν 5, 10, 50, 40 χρόνια. Το σημαντικό είναι να γνωρίζουμε όλε τι αποφάσει tax rulings οι οποίε ισχύουν σήμερα. Αυτή θα είναι και η θέση την οποία θα ε, εκπροσωπήσω στον τριμερή διάλογο, πιστεύω. Πράγματι, κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε μαζί σα ότι είναι πρόοδο για το γεγονό γεγονός ότι ετέθησαν αυτά τα θέματα στο τραπέζι του ΕΚΟΦΗΝ. Αλλά εάν αυτή η συζήτηση δεν είναι δημόσια, γνωρίζουμε ότι η οικονομική και φορολογική πολιτική, μάλλον είναι φορολογική πολιτική, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και ότι υπάρχει κοινοβουλευτικό έλεγχο σε κάθε κράτο μέλο, βεβαίω και ότι οι εκπρόσωποι του λαού καθενό από αυτά τα κράτη έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν την κυβέρνησή του και το φορολογικό καθεστώ που ψηφίζει για του φόρου. Αλλά ε, χάρη σε εσά και χάρη στους συναδέλφους σας στο ΕΚΟΦΗΝ γίνεται μια τέτοια συζήτηση στο εσωτερικό του στο ΕΚΟΦΗΝ και θα θέλαμε αυτή η συζήτηση να είναι πραγματικά δημόσια και προσβάσιμη στους πολίτες. Σας ε, ευχαριστούμε ε, για την παρουσία σας και για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα δύο λεπτών για να ε, συνοδεύσω εκτός της αίθουσας τον Πρόεδρο του ΕΚΟΦΗΝ και να ε, αποδεχτώ και τους προσκεκλισμένους μας. Ευχαριστώ.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

Ευχαριστώ. Messieurs les ministres, mes Κύριε Υπουργέ, συνάδελφοι, άρχεται το δεύτερο τμήμα της συνάντησής μας, της προσωρινής επιτροπής τάξε. Ευχαριστώ τους τέσσερις υπουργούς που είναι εδώ παρόντες και που δέχθηκαν όχι μόνο να έρθουν ενώπιον της Επιτροπής μας, πρεμιέρα είναι αυτή, δεν νομίζω ότι έχει μιλήσει ταυτόχρονα καμία επιτροπή στο Κοινοβούλιο με τέσσερις υπουργού, τόσο σημαντικούς θα τολμούσα να πω στο ΕΚΟΦΗΝ. Μόλις προηγουμένω μίλησε ο Υπουργό κ. Γραμμενιά, θα ακούσουμε και τώρα τον κύριο Παντοάν, Υπουργό της Ιταλίας, Οικονομικών της Ιταλίας, τον κύριο Σαπέν της Γαλλίας, τον Λουίς Δεγκίντος της Ισπανίας και τον Βόρκαμ Σόιμπλε Υπουργό τη Οικονομικών τη Ομοσπονδιακή Γερμανία Γνωστοί και οι τέσσερις, δεν του παρουσιάσω. Θέλω απλώ να υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή, αυτή Επιτροπή δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δώσει μια πολιτική απόφαση στο σκάνδαλο που, που απεκάλυψε ε, οι δημοσιογράφοι, ιδίως το LuxLeaks, για τον τρόπο με τον οποίο ε, ε, φορολογούνται τα κέρδη στα 28 κράτη-μέλη της Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο κάποια, κάποιες σημαντικές πολυεθνικές ε, μπορούν να αποφύγουν να πληρώσουν μεγάλο μέρος των φόρων χρησιμοποιώντας τα πολλά φορολογικά καθεστώτα στην Ένωση ή τα ιδιαίτερα πλονεκτήματα που παρέχει ο νόμος ή οι διοικητικές πρακτικές επιχειρήσεις αυτές μέσα στην Ένωση θα προχωρήσουμε σε μια έρευνα που κρατάει ήδη 6 μήνες και οργανώνουμε απόψε μαζί σας ε, μια τελευταία ανταλλαγή απόψεων δημοσία με υπουργού ε, που έχουν την ευθύνη των οικονομικών. Η έρευνά μας αφορά και τα 28 κράτη-μέλη. Περιμένουμε ακόμα κάποιες απαντήσεις και χαιρόμαστε που τέσσερις από τα σημαντικότερα κράτη-μέλη της Ένωσης επέλεξαν να απαντήσουν όχι μόνο εγγράφως αλλά και να έρθουν οι ίδιοι υπουργοί ενώπιόν μας. Θα τους ακούσουμε καταρχήν και κατόμι θα δώσουμε το λόγο στους εισηγητές και 12 αγορητές όπως και με τον κύριο Γκραμενιά και λόγω της πίεσης του χρόνου θα παρακαλούσα όλους τους αγορητές μέλη της Επιτροπής να τηρήσουν δίλεπτο στην παρέμβασή τους για να μπορέσουν να απαντήσουν στις ε, ερωτήσεις σας οι υπουργοί παρόντες. Καταλαβαίνω ότι έγινε καταμερισμός των αρμοδιτών μεταξύ των προσκεκλημένων και θα μιλήσουν Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Γερμανία. Με συγχωρείτε βόλγκαν, Wolfgang. για πέντε λεπτά. Όχι ότι θα σας χτυπήσω αν ξεπεράσετε το πεντάλεπτο, αλλά καταλαβαίνετε όλοι ότι ο χρόνος πιέζει. Ξεκινά ο κύριος Παντοάν. Και ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι καλησπέρα σα. Πρέπει να σα πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ ε, για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τι ε, φορολογίε και τα φορολογικά συστήματα. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ε, συζήτηση ευρωπαϊκή σχετικά με τη φορολογητέα ύλη αλλά και με τι επιθετικέ φορολογικέ πολιτικέ. Η συζήτηση με την Επιτροπή ΤΑΞ μα προσφέρει μια θαυμάσια ευκαιρία για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα θέματα. Όσον αφορά την Ιταλία, αυτά είναι θέματα πολύ μεγάλη σημασίας. Ε, γνωρίζουμε και ξέρετε και εσείς ότι έχουν καταβληθεί πάρα πολλέ προσπάθειες στο πλαίσιο της BEPS, του G20, του ε, ΟΑΣΕ, αλλά επίσης θέλω να επισημάνω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια εντελεχέστερη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέρυσι, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της ε, Ιταλικής Προεδρίας, ε, εισαγάγαμε μια ιδέα να υπάρχει ένα πίνακα καταρχάς για να μπορεί κανείς εκεί να δει την πρόοδο που επιτυγχάνεται στο θέμα της BEPS. Ε και επίσης συντάξαμε μια ημερήσια διάταξη Ευρωπαϊκής Ένωσης BEPS. Ε η Λετωνική Προεδρία δούλεψε πολύ σκληρά για την εφαρμογή και υλοποίηση αυτού του θεματολογίου. Και το ίδιο κάνει ακριβώς και η Προεδρία του Λουξεμβούργου. Για να μπορέσουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα φαινόμενα BEPS ε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απαραίτητο κατά την άποψή μου να ενισχύσουμε τις ε, προληπτικές δράσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως αναφορά την ε, φορολογία. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε αυτό το θέμα ε, τον Ιανουάριο εγκρίθηκε μία τροποποίηση της οδηγίας ε, για την καταβολή μερισμάτων ε, από τις μητρικές και τις θηγατρικές εταιρείες και εκεί περιλαμβάνεται μία ρήτρα de minimis. Είναι πολύ ικανοποιημένος για το ότι ελπίζω να έχουμε μία επιτυχία στο Συμβούλιο και όσον αφορά την πρόταση τροποποίησης σχετικά με τους κανόνες και τα συμφέροντα. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συζητήθηκε στις 17 του περασμένου Ιουνίου, μια σημαντική πρωτοβουλία την οποία εγκρίνουμε εμείς και στηρίζουμε αποτελεσματικά. Το κείμενο περιγράφει λεπτομερώς τα κενά που υπάρχουν στην νομοθεσία και υπογραμμίζει την ανάγκη μιας ευρείας ε, αναθεώρησης της υφιστάμενης ε, νομοθεσία, προσαρμόζοντάς τη στο παγκοσμιοποιημένο, ψηφιακό και κινητό περιβάλλον του σήμερα. Στην κοινή επιστολή που αποστήλαμε μαζί με τον Μισελ και τον και στον επίτροπο κ. Μοσκοβισή πέρυσι τον Νοέμβριο υπογραμμίσαμε την ανάγκη η Επιτροπή να αναλάβει τις αναγκαίε πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσει τα διάφορα προβλήματα που συνδέονται με τα φαινόμενα BEPS. Θεωρώ ότι η ανακοίνωση και οι πέντε δράσεις κλειδιά είναι μια πρώτη απάντηση στα αιτήματά μας και ευχαριστώ την Επιτροπή για την πρωτοβουλία αυτή. Το πρόγραμμα δράσης που της Επιτροπής έδωσε κεντρικό ρόλο στην ε, στην επανεξέταση της πρώτης οδηγίας σε μια κοινή ενοποιημένη φορολογητέα βάση για τις επιχειρήσεις που είναι μεταρχικά CCCDP. Πρόκειται για μια επιλογή που συμμερίζομαι. Ο καθορισμός κοινών κανόνων για τον καθορισμό της φορολογητέας βάση των επιχειρήσεων θα μείωνε, θα εξάλληφε τη δυνατότητα να, γίνει εκμετάλλευση διαφορών μεταξύ κρατών μελών και φορολογικών ε, δραστηριοτήτων σε κάθε κράτος μέλος. Η διασυνοριακές λοιπόν δραστηριότητε θα κέρδιζαν σημαντικά και από την άποψη της απλοποίησης, τη μείωση της, της διοικητικής επιβάρυνσης και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, παρέχοντας ταυτόχρονα καλύτερο πλαίσιο για την ανάπτυξη και την επένδυση. Στο πλαίσιο αυτό η σταδιακή προσέγγιση, το step by step που προτείνει η Επιτροπή, ε, πρέπει να παροτρινθεί να προχωρήσει. Το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής αντιμετωπίζει και την ανάγκη ε, αντιμετώπισης των αθέμητων φορολογικών πρακτικών και των επιθετικών φορολογικών πρακτικών που ε, δεν μπορούν να λειτουργήσουν μέσα στα πλαίσια μιας ε, ε εξισορρόπησης των φορολογικών, των, φορολογικών, των φορολογικών δραστηριοτήτων και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό σε εθνικό επίπεδο, υπονομεύοντας την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιβλαβής ε, φορολογική, ο επιβλαβής φορολογικός ανταγωνισμός που οδηγεί στη μετακίνηση των επιχειρήσεων και των κερδών από χώρα σε χώρα, φέρει σε κίνδυνο την ικανότητα άλλων των μελών να εισπράξουν τα, τους οφειλόμενους φόρους, μειώνοντας την διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων για την αναδιαμόρφωση της φορολογικής επιβάρυνση ώστε να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα δράση προτείνει την ενίσχυση του ρόλου του, της ομάδας κώδικα διοντολογία για, την επιχείρηση, για φορολογία των επιχειρήσεων, θέμα που και αυτό μας βρίσκει σύμφωνος και πρέπει να συνεχιστεί. Συμπερασματικά έχουμε την συγκεκριμένη δυνατότητα να επιτύχουμε πρόοδο γρήγορα στην αντιμετώπιση φαινομένων BEPS ε και να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συνοχή των φορολογικών συστημάτων μέσα στην Ένωση προς και μειώνοντας τις δυνατότητες υποθετικού φορολογισμού, φορολογικού προγραμματισμού και απλοποιώνοντας ε, την ε, το κόστος των δραστηριοτήτων και, την, και βελτιώνοντας την ασφάλεια δικαίου στην Ένωση. Το Κοινοβούλιο συμβάλλει σημαντικά στις εργασίες του Συμβουλίου και είμαι βέβαιος ότι η συνέχιση του διαλόγου μεταξύ μας που ξεκινά σήμερα θα ενθαρρύνει πολύ συγκεκριμένη ε, δράση και ουσιαστικά αποτελέσματα στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ξεκινήσατε με την παρέμβασή σας σε αυτή τη συζήτηση, ιδίως αναφέροντας την πρωτοβουλία BEPS του ΩΣΑ. Θα δώσω το λόγο στον Υπουργό κύριο Σαπάν της Γαλλίας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που απευθύνατε σε τέσσερις υπουργούς. Θα έλεγα ότι έχει και συμβολική σημασία η παρουσία μας και των τεσσάρων εδώ. Χρειάζεται να παρέμβουμε αποτελεσματικά και γρήγορα στον τομέα αυτών, στη, να καταπολεμήσουμε τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τον επιθετικό φορολογικό προγραμματισμό. Δεν χρειάζεται καν να αναφέρω γιατί τα ανέφερε πολύ σωστά ο συνάδελφος από την Ιταλία. Ο στόχος είναι να μην υπάρχει ένας ε, φορολογικός ανταγωνισμός ε, τόσο μεγάλος μεταξύ των κρατών της Ένωσης. Χρειάζονται όμως και καταπολέμηση του ε, φαινομένου στο παγκόσμιο επίπεδο. Εάν το δούμε στο παγκόσμιο επίπεδο, η κατάσταση δημιουργεί προβλήματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να δικαιολογήσει και να γίνουν αποδεκτά από την κοινή γνώμη. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν η Γαλλία θεωρεί ότι πρέπει συλλογικά να αποφασίσουμε τους κανόνες του παιχνιδιού έτσι ώστε να περιοριστεί αυτή η δυσμενής για όλα τα κράτη χρήση του φορολογικού προγραμματισμού για να είναι ξεκάθαροι οι κανόνες του ανταγωνισμού. Ε, από το 2014 ξεκίνησαν από την πλευρά της Επιτροπής μια σειρά προτάσεων ε, το Μαΐου 2014 έγινε η πρώτη πρόταση για την οδηγία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από τις φορολογικές διοικήσεις. Είναι μια σωστή πρωτοβουλία την οποία την υποστηρίζει η Γαλλία και ε, το 2015, από το 2015. Ξεκίνησε ένα πρόγραμμα δράσης, η κατάρτιση μιας ε, προγράμματος δράσης που θα ε, δημιουργήσει ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα συνολικά και η Γαλλία επίσης υποστηρίζει αυτή την πρωτοβουλία. Εγώ θα ήθελα να σταθώ περισσότερο όμως σε κάποιο άλλα συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή, τον ελάχιστη φορολογιατό αρχή de minimis. Κάτι που συζητήθηκε στη, στο Συμβούλιο του, στο Λουξεμβουργό πριν από λίγες εβδομάδες το ευρωπαϊκό δίκαιο μπορεί να ασχολήθηκε μάλλον μέχρι τώρα στην αποφυγή της διπλής φορολόγησης. Και αυτό ήταν απαραίτητο. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να φροντίσουμε πλέον να γίνεται είναι να πάμε ένα βήμα παραπέρα και να φροντίσουμε ότι οποιοδήποτε εισόδημα θα φορολογείται τουλάχιστον μία φορά και σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό. Αυτό είναι η αρχή που θα πρέπει να εισαχθεί τώρα πλέον στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο γιατί είναι κάτι που δεν συμβαίνει ακόμα. Και αν κάτι τέτοιο τελικά νομοθετηθεί θα, έχουμε, ε, θα πάψουν αυτές τις τρευλώσεις του ανταγωνισμού που δημιουργούν τόσα προβλήματα στην ενιαία αγορά. Το ζήτημα αυτό συζητείται στο πλαίσιο του Συμβουλίου, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Συμβουλίας για τους στόχους και τα δικαιώματα του 2013. Συμφωνώ με τις απόψεις που έχει εκφράσει η Επιτροπή στις 17 Ιουνίου 2015 στην ανακοίνωση της για το θέμα αυτό. Και η πρώτη μας ευκαιρία ε, ε, να αναλάβει δράση Συμβούλιο, για το θέμα αυτό το Συμβούλιο είναι αυτή η οδηγία η οποία αναφέρθηκε για τις ε, σχέσεις ε, των ε, μητρικών θηγατρικών εταιριών. Κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνεται εάν αυτή τη στιγμή το ένα κράτος μέλος αποφασίσει να μην φορολογήσει τα κέρδη μιας εταιρείας δεν υπάρχει ε, κάποιο, σύστημα το οποίο θα φροντίσει ε, τουλάχιστον κατελάχιστον να φορολογηθούν ε, αυτά τα κέρδη κάπου. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να δημιουργηθεί έτσι ώστε τα, τα, τα, οποιοδήποτε εισόδημα, οποιοδήποτε κέρδο να φορολογείται τουλάχιστον μία φορά στο έδαφο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα πρέπει, παρόλο που είναι άλλο ζήτημα, να επιδιώξουμε την εναρμόνιση μακροπρόθεσμα των φορολογικών συστημάτων. Βεβαίω γνωρίζετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ε, χρειάζεται ομοφωνία. Αλλά ε, η εισαγωγή στο ευρωπαϊκό δίκαιο της αρχής της αποτελεσματικής φορολόγησης είναι ένα σημαντικό βήμα αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην συγχαίουμε την εισαγωγή αυτή τη αρχή με την πλήρη αναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων. Γιατί φοβάμαι ότι κάποιοι θα προσπαθήσουν να, κάνουν αυτή, ε, τη, τη, να, να βλέξουν αυτά τα δύο συζητήματα έτσι ώστε να μην προχωρήσουμε σε κανένα από τα δύο. Καλωσορίζουμε λοιπόν τι νέε πρωτοβουλίε τη Επιτροπή γνωρίζοντα ότι δεν μπορούμε παρά να προχωρήσουμε βήμα-βήμα ε, πηγαίνοντα προ την εναρμόνιση. Αυτή τη στιγμή είναι. Ε, ε, προαιρετικό να, κινηθεί, ε, να κινηθούν τα κράτη-μέλη προς την εναρμόνιση, ωστόσο μια τέτοια ε, εναρμόνιση θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Η Γαλλία υποστηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες και θα συμμετάσχει ενεργά στη συζήτηση. Αυτά, αυτές τις θέσεις ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, τονίζοντας τα κυριότερα σημεία που αποσχολούν τη χώρα μου και σας ευχαριστώ για την, πρόσκληση, για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε ε, Υπουργέ. Θα δώσω το λόγο στον Υπουργό ε, Λουίς Τεγκίντος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε, Αντιπρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, ευχαριστώ που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω στην Επιτροπή σας. Είναι μια ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας και με τους αδέλφους για τη φορολογία στην Ευρώπη. Ένα θέμα που έγινε ένας από τους βασικούς στόχους της ε, ημερήσιες θεματολογίες στην Ευρώπη που πρέπει να συνεχίσουμε να υλοποιούμε αν θέλουμε να εμβαθύνουμε την ενιαία αγορά. Όπως ξέρετε, ο συντονισμός των φορολογικών πολιτικών του κατωμερών απαιτεί πολλά πράγματα, διότι υπάρχουν εμπόδια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε μειονεκτική κατάσταση σε σχέση με τις συμμεταπές επιχειρήσεις όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό. Η ίσπραξη κατόπιν είναι δεύτερο θέμα οι, φορολογι... οι επιθετικές φορολογικές δραστηριότητες και δημιουργούν αθέμητα κέρδη, κάτι που είναι σημαντικό γιατί υπονομεύει την αρχή της διαφάνειας που είναι βασικό σε όλα τα φορολογικά συστήματα σε, σε δημοκρατικές χώρες ενώ σε ευαίσθητες ιδιαίτερα εποχές όταν όλοι καταβάλουμε προσπάθειες ε, βελτίωσης των δημοσίων οικονομικών βλάπτει τα τελευταία. Γι' αυτό εμείς υποστηρίζουμε τις αρχές της ε, Φορολογική δικαιοσύνη μεταξύ πληρωμή, συζητώντα μια ισορροπία μεταξύ πληρωμή φόρων και ισοτιμία. Τώρα, η κατάχρηση των λεγόμενων tax rulings είναι θέμα συζήτηση στην Ευρώπη. Ε, Δημιουργούν, ε, οι δυνατότητε αυτέ μπορούν να είναι εργαλεία σε κάποιε περιπτώσει θετικά γιατί βοηθούν τι επιχειρήσει, Ωστόσο, σε πολλέ χώρε όπω γνωρίζετε, χρησιμοποιούνται τα tax rulings ε, με κακή προαίρεση, δημιουργώντας αθέμητο φορολογικό ανταγωνισμό, κάτι ε, που είναι απαράδεκτο σε κράτη που μετέχουν σε μια πολιτική ένωση. Η Ισπανία θεωρεί ότι η συνεργασία είναι αναγκαία μεταξύ όλων και η χώρα μου συνεργάστηκε πλήρως ε, στον τομέα αυτό και αυτό συμβαίνει και με άλλε χώρε. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η ενίσχυση της συνεργασίας και της διαφάνειας στην Ένωση είναι βασική προϋπόθεση για να εμβαθύνουμε την ενιαία αγορά. Όσα έχει υποβάλει στον τομέα αυτό μια σειρά προτάσεων όπως την, τον έλεγχο, ε, το BEPS, ε, την, το Συμβούλιο υιοθέτησε την περσμένη εβδομάδα τις εκθέσεις για τις 15 γραμμές, ε, καθοδητήρες γραμμές που θα υιοθετήσουμε σύντομα. Η ενημέρωση αναχώρα είναι σημαντική διότι πρέπει, επιτρέπει στις πολυεθνικές να παρέχουν πληροφορίες και στα κράτη να ζητούν πληροφορίες. Οι φορολογικές αρχές μπορούν να, να ανταλλάσσουν πληροφορίες με αντίστοιχες δομές σε άλλες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει ε, την ίδια απέτηση από τις επιχειρήσεις ε, του εξωτερικού που αυτές που έχει και στην, τις δικές της. Χρειάζεται ταυτόχρονα μεγαλύτερο συντονισμός μεταξύ των εθνικών αρχών. Το πρόγραμμα δράσης που παρουσίασε η Επιτροπή πρόσφατα αποτελεί μια εξαιρετική συμβολή στη συζήτηση αυτή, καθώς και η τροποποίηση της οδηγίας για τη διοικητική συνεργασία που αποτελεί ένα πρώτο βήμα για μεγαλύτερη διαφάνεια στην Ένωση. Μετά από πολλά έτη δουλειά πρέπει να τονίσουμε ότι η Ένωση βρίσκεται στη φάση ξεκινήματο μια νέων προτύπων και απαιτήσεων για τη μεταφορά δομένων. Η Ισπανία, το πιτέψω να το πω, ήταν μεταξύ των πρωτοπόρων στην καταπολέμησή τη φοροδιαφυγή. μαζί με την Ιταλία, τη Γαλλία, την Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ξεκινήσει την, την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών αποφάσεων ήδη από το, που θα ξεκινήσει να λειτουργεί από το 2017. Ταυτόχρονα υιοθετήσαμε μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση τη διάβρωσης τη φορολογική βάση των ε, πολιτών, τονίζοντα ταυτόχρονα ότι έφυγαν, καταργήθηκαν μια σειρά ε, φορολογικών δυνατοτήτων όπως οι περιορισμοί για τις δαπάνες ε, των επιχειρήσεων για την, για την υπερχρέωση βασίδιων πόρων κλπ. Ταυτόχρονα, τον επόμενο χρόνο υιοθετούμε με ένα χρόνο νωρίτερα τις διατάξεις για την νομοθεσία για τις ε, κεφαλαϊκές εταιρείες, ούτως ώστε αυτή τη στιγμή η, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων είναι συνυπεύθυνα για φορολογικές απάτες ή φοροδιαφυγή. Ταυτόχρονα έχουμε υιοθετήσει σημαντικά βήματα όπως τη δημοσιοποίηση καταλόγου κάποιων ε, ενόχων καθώς και τη δημοσιοποίηση των φορολογικών καταδικαστικών αποφάσεων. Σύντομα θα τροποποιήσουμε το φορολογικό καθεστώς των, διπλωμά... των ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Κλείνω. Η Ισπανία, όπως σας είπα κυρίε και κύριοι, θέλει να χτυπήσει την, την φοροδιαφυγή και τις αθέμητες φορολογικές πρακτικές. Ως κράτος έχουμε προχωρήσει μια σειρά θεμάτων που έχουμε προωθήσει μια σειρά θεμάτων που, σε, που υιοθετήθηκαν σε διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει τη μάχη κατά των πρακτικών αυτών. Σε μια φάση, σε μια στιγμή όπου προσπαθούμε να, ενσωματώ, να ενοποιήσουμε περισσότερο την Ευρωζώνη, η φορολογική, ο φορολογικό ανταγωνισμό θα πρέπει να γίνει θεμητό και να επιτρέψει να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πραγματικά ενιαίο χώρο. Ευχαριστώ πολύ. Muchas gracias, Luis. Et enfin, la parole à Wolfgang Το λόγο λοιπόν έχει ο Υπουργό Οικονομικών τη Γερμανία, ο κύριο Σόιμπλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Γερμανία χαιρετίζει τι εργασίε αυτή τη επιτροπή, διότι εμεί πιστεύουμε ότι οι φορολογικέ αποφάσει, τα περίφημα tax rulings, δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ω εργαλείο ανταγωνισμού. Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε την ε, αλλαγή της οδηγίας ε, περί ε, αρρωγής στις περιπτώσεις αυτές. Χρειαζόμαστε όμως και εσωτερικά κριτήρια για τις φορολογικές αποφάσεις. Αν δούμε τα BEPS στο σύνολό τους, όπως ακριβώς περιγράφηκαν από το συνάδελφό μου, και αν θέλουμε να ενισχύσουμε τα BEPS, τότε πρέπει από κοινού να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία και το κάναμε ήδη αυτό, άρα δηλαδή είναι θέμα αξιοπιστίας. Να προχωρήσουμε εμείς, Ευρωπαίοι, όλοι από κοινού, και αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε σαφώς ενίσχυση της ομάδας Code of Conduct, του κώδικα διοντολογίας, επί της οποίας θα μου επιτρέψετε να κάνω εγώ κάποιες εισαγωγικέ παρατηρήσεις. Τα έχουμε συμφωνήσει εξάλλου μεταξύ μας. Αυτή η ομάδα είχε ήδη συσταθεί το 1979, διότι ε, ο ανταγωνισμός που υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει χρειάζεται ένα πλαίσιο, πλαίσιο λειτουργίας, να εντάσσεται μέσα σε αυτόν. Τότε λοιπόν όλοι πιστεύαμε ότι οι διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές δεν παραβιάζουν την αρχή του θεμητού και υγιούς ανταγωνισμού. Εν τω μεταξύ βέβαια καταλήξαμε στο ότι δεν μπορούμε αυτό να το αφήσουμε απαράλλαχτο. Καταλήξαμε στο ότι χρειαζόμαστε ελάχιστους φορολογικούς συντελεστέ. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Με βάση το πρωτογενέ δίκαιο οι αποφάσει λαμβάνονται όλες ομόφωνα και αυτό πρέπει κανείς να το έχει κατά νου οποτεδήποτε ασχολείται με τέτοιου είδου θέματα. Αυτή λοιπόν η ομάδα, η ομάδα Code of Conduct δούλεψε τη δεκαετία του 80 κάτω από αυτέ τι παραδοχέ, δούλεψε πάρα πολύ καλά, προσέφερε μία σειρά κινήτρων και η ομάδα αυτή συνέβαλε στο να ε, θεσπιστούν μία σειρά ε, φορολογικών κανόνων οι οποίοι προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές εξελίξεις. Εν τω μεταξύ όμως διαπιστώθηκε ότι χρειαζόμαστε νέα κίνητρα. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να συζητήσουμε για τα κριτήρια του αθέμητου ανταγωνισμού, άρα δηλαδή και για την εντολή που έχει δοθεί σε αυτή την ομάδα και ενδεχομένως να τροποποιηθεί η εντολή. Εν τω μεταξύ νομίζω ότι έχει φτάσει η χρονική στιγμή η ομάδα αυτή να αποκτήσει ένα νέο πρόγραμμα εργασίας και να γίνεται και λόγος για τις περίφημες outbound payments. Αυτό σε σχέση με τις ε, εμβάσματα σε φορολογικούς παραδείσους. Αυτό δεν είναι σαφώς προς όφελος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, εύκολα λέγεται, δύσκολα γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, όμως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Χρειαζόμαστε επίσης ε, αλλαγές στη διαδικασία λειτουργίας της ομάδας. Ε, χρειαζόμαστε αποτελεσματική λογοδοσία της ομάδας τους Υπουργού Οικονομικών. Εμείς οι ίδιοι, οι Υπουργοί Οικονομικών, οφείλουμε να ασχολούμεθα στο ΕΚΟΦΗΝ με τα θέματα αυτά και δεν επιτρέπεται να παραπέμπουμε όλα τα θέματα σε επίπεδο τεχνοκρατικό. Όχι, πρέπει να επιλαμβανόμαστε κι εμεί αυτών των θεμάτων. Βεβαίω θα ήταν πολύ καλύτερα να μην η αρχή της ομοφωνίας αλλά της πλειοψηφίας στην ομάδα γιατί κάτι τέτοιο θα επιτάχυνε τις διαδικασίες. Και επίσης και η λογοδοσία στο ΕΚΟΦΗΝ και αυτή δεν πρέπει να δίδεται απαραίτητα με ομοφωνία να υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία αυτό δεν θα αλλάξει τίποτα αυτά έτσι κι αλλιώς προβλέπονται στο Ευρωπαϊκό Πρωτογενές Δίκαιο και δεν αποτελούν παραβίαση του δικαίου αυτού. Εάν δεν υπάρχει λοιπόν αποτελεσματική παρουσία των θεμάτων στο ΕΚΟΦΗΝ, η ομάδα δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική. Η ομάδα αυτή δεν έχει νομική νομιμοποίηση, αλλά ανταυτού η ομάδα θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει κάποιες νομοθετικές πράξεις και με το περίφημο soft law, τις μη δεσμευτικέ νομικές προτάσεις που παρόλα αυτά καταθέτει, μπορεί όμως να πετύχει πάρα πολλά, μπορεί να προωθήσει κανονισμούς, να οδηγήσει στην εφαρμογή τους η ομάδα στην οποία αναφέρομαι συζητάει μέχρι τέλος του έτους να έχουν τροποποιηθεί οι κανόνες. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι με την ομάδα αυτή και κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες έχουμε στα χέρια μας ένα αποτελεσματικό εργαλείο για να προσφέρουμε περαιτέρω κίνητρα και για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την φόρο διαφυγή αλλά και τον, την αθέμετη εκμετάλλευση φορολογικών διαφορών που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια καταφέραμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολλά, με συγχωρείτε, τώρα όμως δεν έχουμε φτάσει στο τέλος του δρόμου. Οφείλουμε να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά, ακριβώς όπως το κάναμε και με τα tax rulings και με την ανταλλαγή πληροφοριών. Υπάρχουν σχετικές οδηγίες περί επιτοκίων και τα σύναφη. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θεωρώ ότι οι εργασίες της ομάδας Code of Conduct πρέπει να βελτιωθούν και να ενισχυθούν περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ αγαπητέ Βόλφκαν κύριε Υπουργέ. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στους συναδέλφους. Θα ήθελα να τηρήσουμε το χρόνο δύο λεπτά ο κάθε μιλητής Μπορείτε να θαυμάσετε πόσο τήρησαν το χρόνο τους οι υπουργοί, επομένω έδωσαν το παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και εμείς οι βουλευτές. Δεν είναι. Λοιπόν, ε, για να διευκολύνουμε και τη συζήτηση μετά, θα ήθελα να συζητήσω σε ποιον ε, υπουργό απευθύνεστε, αν απευθύνετε μια ερώτηση σε κάποιον συγκεκριμένα. Ξεκινώ ε, με τους συζητητές φυσικά, πρώτα απ' όλα η Ελίσσα. Για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργή. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι δεν υπάρχει καθόλου ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και του Λουξεμβούργου ή των κατοχωρών. Παρόλα αυτά, από το 1997 υπήρχε το νομικό πλαίσιο που επέτρεπε να ζητηθούν πληροφορίες. Γιατί συνέβη λοιπόν αυτό. Μιας και όλοι συμφωνείτε ότι αυτά τα προβλήματα από τις φοροαποφυγής δημιουργούν τεράστια προβλήματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Το δεύτερο μου ερώτημα είναι σε εσά που είστε οι πλέον ισχυροί πολιτικά και οικονομικά ηγέτες της Ένωσης. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι με την παρουσίαση που κάνατε θα υπάρξει μεγαλύτερο συντονισμό στα φορολογικά ζητήματα και θα σημειωθεί πρόοδος. Και αν τα καταφέρουμε θα πρέπει να σας συγχαρούμε. Αν δεν τα καταφέρετε όμως εσείς θα αναλάβετε και την ευθύνη. Τρίτον, υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα στην ημερησία διάταξη, ένα από τα οποία είναι οι συστάσεις αναχώρα, οι εκθέσεις αναχώρα το βρίσκεται στο στάδιο του τριμερούς διαλόγου, αλλά η στάση του Συμβουλίου δεν είναι ενθαρρυντική. Είναι ένα ζήτημα διαφάνειας αυτές οι εκθέσεις αναχώρα, κάτι που το αναφέρατε κι εσείς, ότι είναι ψηλά στι προτεραιότητε σας. Ακούσαμε λοιπόν ότι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία ε, μπλοκάρουν τις διαπραγματεύσεις. Ισχύει αυτό. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες. Πώς θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν σημειώνεται πρόοδος και ποια χώρα από εκείνες του Συμβουλίου μπλοκάρει την πρόοδο. Συζητώντας μετά πέρα από ε, το, το, τον, ε, τον κώδικα διοντολογίας, πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα, γιατί δεν, αρκούν αυτά τα εργαλεία. Βρισκόμαστε σε μια ενιαία αγορά και χρειάζεται να υπάρξει πολύ μεγαλύτερο συντονισμός και συνεργασία στα θέματα τα φορολογικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ελίζα. Και θα δώσω το λόγο στον δεύτερο συνεισηγητή, Μίκαρ Τόερετ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και για το γεγονός ότι μπορέσατε να πείσετε τους υπουργούς να έρθουν εδώ. Και σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργή, είναι πολύ σημαντικό που ήρθατε. Εμείς ε, ως εισηγητές ε, αναζητήσαμε τη νέα ποιότητα που έχει προκύψει από το σκάνδαλο LuxLeaks. Ε, το γεγονός ότι υπάρχει φορά φυγή, το ξέραμε όλοι, αλλά το γεγονός ότι χάνονται εκατοντάδες εκατομμύρια, αυτό δεν το γνωρίζαμε. Ε, διαπιστώσαμε λοιπόν ότι τα εθνικά πολύ περίπλοκα εθνικά φορολογικά συστήματα ε, προκαλούν αυτά τα παραθυράκια από τα οποία χάνονται όλα αυτά τα εκατομμύρια. Και το ερώτημά μου είναι το εξή. Από ό,τι φαίνεται ε, σε, στο ΕΚΟΦΗΝ και κλεισμένο των θυρών τα συζητάτε αυτά πάρα πολλά χρόνια. Και τι γίνεται τελικά, πού βρίσκεται η πολιτική αντίδραση. Εμείς οι απλοί πολίτες διαρωτώμεθα γιατί όλη αυτή η μυστικοπάθεια. Μήπως μπορείτε και εμείς ε, να μας πείτε λιγάκι ποιος αντίδρα, πού υπάρχει το πρόβλημα. Γιατί νομίζω Νομίζω ότι είναι σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εμπόδισε τα κράτη-μέλη, ούτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για μας εντωμεταξύ είναι απόλυτα σαφές ότι χρειαζόμαστε ένα ελάχιστο πλαίσιο, μια ελάχιστη κοινή φορολογική βάση για να μην υπάρχει ανταγωνισμός μέσα από τους συντελεστές. Και εδώ πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ε, Κύριε Σόιμπλε, απευθύνομαι σε εσά ε, ω ε, συμπολίτη σα. Η Γερμανία, το Bundesrat συγκεκριμένα, δεν συμφωνεί με τι προτάσει Κομισιόν. Τοποθετήθηκε αρνητικά. Ε, Επίση, τίθεται το ερώτημα κατά πόσον σύμφωνα με το άρθρο 89 και σύμφωνα με το άρθρο 88 κατά πόσον ε, αυτές οι δύο παράγραφοι καλύπτονται από τα tax rulings. Δηλαδή, συμφωνείτε τι είναι αυτά τα tax rulings, συμφωνείτε όλοι σας ε, και γιατί τελικά δεν συμφωνούμε να υπάρξει ένας ε, διαιτητικός φορέας, ένας διαιτητικός οργανισμός. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, τον θεωρούμε αυτό απολύτως απαραίτητο. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Πάμπλο από το από το ΕΛΚ. Εδώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη κύριε Υπουργή, σας ευχαριστούμε για την ε, παρουσίαση στην συνάντηση της Επιτροπής μας. Αυτό που αποκάλυψαν τα LuxLeaks, νομίζω, είναι ότι μας έδειξαν με ε, δεδομένα και με στοιχεία ότι χρειαζόμαστε μια πραγματική ένωση οικονομική ε, και φορολογική τελικά και θα μας δώσουν την όθηση που χρειάζεται για να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση αυτές οι αποκαλύψεις και οι οι προτάσεις που ακούμε ακούγονται πολύ φιλόδοξες. Από την πλευρά της η Επιτροπή έχει επίσης καταθέσει ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο δράσης. Το ερώτημά μου όμως είναι το εξής. Πότε αναμένεται ε, να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα τελικά. Πότε πιστεύετε εσείς ότι θα υλοποιηθούν. Πότε μπορούμε να εγγυηθούμε στους πολίτες μας ότι αυτά τα προβλήματα δεν θα ξαναεμφανιστούν. Σταματήσουν. Μια άλλη ανομαλία, περίεργη κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η κατάσταση με το Γιβραλτάρ. Και φοβάμαι ότι θα πρέπει να το, να το αντιμετωπίσουμε και αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να το παραμερίσουμε. Και θα ήθελα να γνωρίσω, να γνωρίσω ποια είναι η θέση σας, όλων σας και ιδιαίτερα του κ. Ντεγκίνητο για το θέμα του Γιβραλτάρ. Σα ευχαριστούμε από τους σοσιαλιστές. Κύριε Σίμων, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι εργασίες εδώ κατέδειξαν ότι υπάρχει και η κρατικά οργανωμένη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή και όχι μόνο τα παρατηράκια. Υπάρχει εδώ κρατικά οργανωμένη φοροαποφυγή και μάλιστα αυτά τα κράτη κερδίζουν από τους φόρους και κερδίζουν και οι ε, μεγάλες πολυεθνικές όχι όμως οι μικρομεσαίες. Έχουμε την έκθεση Νίντεμάε με την οποία κάναμε μία μελέτη. Διαπιστώθηκε ότι 50 μέχρι 70 δις το χρόνο χάνονται ως φορολογικά έσοδα οποτεδήποτε προκύπτουν τέτοιου είδους διαδικασίες. Και προσθέτεται και άλλα πάρα πολλά. Μιλάμε δηλαδή για το ίμιση του ενωσιακού ε, προϋπολογισμού ε, και επίσης, και επίσης ένα μεγάλο ποσό του προϋπολογισμού της ε, Ομοσπονδιακής Γερμανίας. Βλέποντας λοιπόν όλα αυτά, εντυπωσιάζει πάρα πολύ το ότι η συζήτηση τα τελευταία χρόνια ήταν απλά επιφυλακτική. Αν δούμε άλλα προβλήματα στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι η σημασία αποδίδεται σε κράτη-μέλη τα οποία αισθάνονται σε μειονεκτική θέση. Πολλοί λοιπόν ομιλούν για ανοχή. Ανοχή και αυτό νομίζω ότι και άλλοι θέλουν να το θέσουν το ερώτημα και σας ερωτώ γιατί θεωρείτε εσεί ότι το πρόβλημα έλαβε τόσο τεράστιο διαστάσεις. Ε, η ε, συζήτηση, η πολιτική δεν έχει γίνει ακόμα δημόσια. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο όσον αφορά την φορολογική βάση ε, και του εταιρικού φόρου. Το βρίσκω πάρα πολύ καλό ότι θα κατατεθεί πρόταση, αλλά η πρόταση αυτή θα περιοριστεί σε φορολογική βάση κοινού φόρου επιχειρήσεων χωρίς ενοποίηση. Εσείς λοιπόν είσαστε πρόθυμοι να ενοποιήσετε και να ομογενοποιήσετε αυτό το φόρο στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρχει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Σε ευχαριστώ Πίτερ για το ECR, ο Αντιπρόεδρος Μπερν Λούκε. Το ερώτημά μου αφορά εσάς ε, κύριε Σόιμπλε. Θα συμφωνούμε όλοι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μεγάλο σκάνδαλο. Μάθαμε για εταιρείε ε, οι οποίες ε, προτίθενται να μειώσουν τη φορολογία των κερδών τους σε κάτω από 1%. Μιλάμε για δισεκατομμύρια τα οποία χάνουν τα δημόσια ταμεία. Και το πρώτο μου ερώτημα προς εσάς είναι το εξής. Έχουν περάσει δέκα μήνες από τότε που πρωτοξέσπασε το σκάνδαλο. Έχετε υπολογίσει άραγε πόσα δις έχασε η Γερμανία με τη μορφή των φορολογικών εσόδων και μπορείτε να μας ανακοινώσετε το ποσό αυτό. Πρώτο ερώτημα ήταν αυτό και περνάω στο δεύτερο. Είναι δύσκολο να βρει κανείς ευρωπαϊκές λύσεις. Εδώ σε αυτή την επιτροπή δουλεύουμε επί του θέματος, το κάνουν και άλλοι ε, φορείς. Αναφερθήκατε στην αρχή της ομοφωνίας. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορούν να επιτευχθούν πάρα πολλά ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της ομοφωνίας. Όμως σε εθνικό ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί κανείς να κάνει κάτι. Εσείς πιστεύετε ας πούμε ότι στη Γερμανία μέσω της ε, νομοθεσίας ή με άλλες διαδικασίες ε, μπορούν οι φορολογικές αρχές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη φοροαποφυγή που δημοσιοποιήθηκε μέσω του σκανδάλου LuxLeaks. Και άλλη ερώτηση. Εσείς συγκεκριμένα ως Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας τι ακριβώς κάνατε έτσι ώστε η φοροαποφυγή να αντιμετωπιστεί μέσα από εθνικε πρωτοβουλίες. Και αν δεν κάνατε τίποτα, αν όχι δηλαδή, γιατί πιστεύετε ότι σε εθνικό επίπεδο δεν πρέπει κανείς να κάνει τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Μπέρντ. Για τους φιλελεύθερους, η κόρα. Okay, uh, thank uh, Ευχαριστώ που ήρθατε. Μία ερώτηση προς τον κύριο Σαππάν. Η πρακτική Ποιος είναι, κατά την άποψή σας, ε, ο ρόλος των ε, εταιριών έρευνας και ανάπτυξης και της γαλλικής κυβέρνησης στην ε, φοροαποφυγή της εφημερίδες, κάποια άρθρα που λένε ότι θέλετε να προωθήσετε την έρευνα και την ανάπτυξη στην Γαλλία εις βάρος άλλων κρατών μελών. Προς τον κύριο Σόιμπλε, ποια είναι η άποψή σας για το ότι πολλά κράτη-μέλη δεν απάντησαν στα αιτήματα της Επιτροπής μας ε, για τα tax rulings, μεταξύ αυτών και η Γερμανία. Τι άποψη έχετε περί αυτού αν ε, λάβετε υπόψη το, την έκκληση πολλών κρατών μελών να βελτιωθεί το tax ruling στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την έκθεση των ε, LuxLeaks. Ευχαριστώ Κόρα. Η Παλώμα Λόπες για την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους υπουργούς που ήρθαν εδώ τέτοια ώρα. Μετά το LuxLeaks δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μια συνένεση προς τα κάτω διότι αυτό θα είναι μια συλλογική αποτυχία. Θα ήταν καλό να υπάρξουν συμφωνίες που θα πηγαίνουν στην αναγκαία εναρμόνιση σε φορολογικό επίπεδο στην φορολογία επιχειρήσεων, την καταβολή των φόρων στις χώρες όπου εισπράττονται τα, ε, τα κέρδη και μια σειρά άλλων μέτρων που θα απέφευγε όχι μόνο θεωρητικά αλλά και στην ουσία ε, την, μιας κατάστασης όπου η πραγματική οικονομία και πρακτική θα εμποδίζουν το φορολογικό dumping και την φοροαποφυγή που είναι προς όφελος των πολυεθνικών, των μεγάλων τραπεζών και συγκεκριμένων επενδυτών ενώ ταυτόχρονα πλήττουν τους εργαζόμενους και τον πληθυσμό να, να υποβάλλονται σε μεγάλη βαριά φορολογία. Ταυτόχρονα θα έδινε περισσότερους πόρους στο, στο δημόσιο για να τα επενδύσει στην ανάπτυξη της Ευρώπης. Για να προχωρήσουμε πρέπει να μιλήσουμε και για διαφάνεια. Απευθύνομαι προς τον κύριο Ιντεγκίντος για το θέμα αυτό. Μιλήσατε για τη διάσταση της διαφάνειας. Ωστόσο, αντιταθήκατε στο Συμβούλιο από ό,τι φαίνεται σε μια μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια όπως απαιτείται από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αντίθεσή σας αυτή δυστυχώς δεν είναι έκπληξη, τουλάχιστον ε, για μένα, διότι έχετε εγκρίνει φορολογική αμνηστία που, με, την οποία, με δεν συμφωνώ, που ενώ επιβάλλατε συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας με, σε περιοχές Φορολογική ευκολίας μόνο και μόνο για το σκοπό αυτό. Πρέπει να θυμίσουμε ότι η φορολογική διαφάνεια είναι βασική δημοκρατική επιταγή. Πρέπει να σεβαστούμε, να καταλάβουμε ότι φορολογική διαφάνεια δεν σημαίνει μόνο να παρέχουμε στατιστικά δεδομένα. Ευχαριστώ Παλώμα. Για τους πράσινους, η Εύα Ζολή, αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους Υπουργούς ε, για την παρουσία τους εδώ μαζί μας τέσσερις χώρες οι οποίες θεωρούνται θύματα της ύπαρξης των φορολογικών παραδείσων. Και αναρωτιέται κανείς γιατί αυτές οι χώρες που εκπροσωπούνται εδώ δεν ανέλαβαν πρωτοβουλία πιο νωρί και με μεγαλύτερη ένταση. Κύριε Σόιμπλε, ε, μιλήσατε για την ομάδα του κώδικα βιοντολογίας ε, και την έκθεση του την αποστήλατε την μοιραστήκατε με το Bundestag, με το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Γιατί δεν την μοιράζεστε και με την Επιτροπή Τάξ σε αυτό εδώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Σαπά, η Γαλλία μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια χώρα που βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος, ε, τη αγώνα κατά του σφοροαποφυγής. Ε, Αλλά αποφασίζετε να δημιουργήσετε αυτές τις, τους ειδικό φορολογικό καθεστώς για τις εταιρείε έρευνας και ανάπτυξης ενώ γνωρίζουμε ότι εκατομμύρια θα ε, χαθούν από το φορολογική βάση τη γαλλική μέσω αυτού του συστήματος. Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί η εισαγωγή αυτού του μέτρου που ενισχύει αυτόν τον ε, αέναο κύκλο, τον φαύλο κύκλο. Κύριε Δικίντος, και εσείς μιλήσατε κατά των φοροαποφυγής, αλλά ψηφίσατε νομοθεσία η οποία επιτρέπει ε, στις τράπεζες ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς το οποίο τους επιτρέπει να αυξήσουν τα κέρδη τους ακόμα περισσότερο. Υπάρχει συνοχή. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι δεν εργάζεστε πια ούτε για την PricewaterhouseCoopers ούτε για τους Lehman Brothers. Ο Αντουάν Τελτούρ είναι η πέτρα του σκανδάλου, ήταν αυτό που μα άνοιξε τα μάτια με το LuxLeaks. Αλλά είναι ο μόνο μαζί με τον Έντουαρτ ε, παρά να ε, απειλείται με φυλάκιση, επειδή είναι ο μόνο ο οποίο μα δημοσιοποίησε, μα έδωσε αυτά τα στοιχεία και δεν τον προστατεύει, δεν τον προστάτευσε κανεί. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα μόνο να συζητήσω να αποφύγουμε τις προσωπικού χαρακτήρα παρατηρήσεις. Για την ομάδα EFTD, Μάρκο Βάλλη. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ και τους υπουργούς για την παρουσία τους. Άκουσα τις παρατηρήσεις τους ε, και δηλώσεις τους που πηγαίνουν προς μια κοινή κατεύθυνση με πεποίθηση μάχης κατά της φοροδιαφυγής και δροφογής. Ωστόσο, στην Ιταλία προσπαθώ εδώ και καιρό να εξηγήσω στους ε, ε, Ιταλούς μικρομεσαίους επιχειρηματίες που πεθαίνουν ε, κυριολεκτικά γιατί κάποιοι αυτοκτονούν από τους πολλούς φόρους να μην μετακινούν τις επιχειρήσεις τους κάτι που θέλουν γιατί δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις μεγάλες πολυεθνικές που μπαίνουν στα Υπουργεία της Οικονομίας όπως βλέπουμε σε διάφορες χώρες, υπογράφουν συμφωνίες με τις χώρες εκείνες και περνούν μια χαρά πληρώνοντας συχνά φόρο κάτω από 1%. Προσπαθώ να τους εξηγήσω λοιπόν αυτή την κατάσταση ότι κάνουμε κάτι και θα τους πω ότι ήρθαν εδώ οι Υπουργοί Οικονομικών, πρέπει να ξυπνήσετε δεν υπάρχει χρόνος να χάσουμε. Ήρθε στην Ολομέλεια ο Γιούνκερ και μας είπε ότι δεν υπάρχει Ένωση, δεν υπάρχει Ευρώπη. Τι έχει η Ευρώπη. Ευρώ, λιτότητα, 150 δις προϋπολογισμών ε, που είναι κύριος πελατειακού χαρακτήρα κρατών και κομμάτων και ένα σχέδιο και μέσα σε όλα αυτά το, η φορολογική εναρμόνιση κάπου χάθηκε προσπαθώντας ε, να... Όλα αυτά οδηγούν σε αύξηση του ευρωσκεπτικισμού που... σε όλες τις χώρες, γιατί δεν προχωρά η Ευρώπη. Έχετε πρόθεση να κάνετε κάτι, είπε και η συνάδελφος προηγουμένως ε, η... στη συζήτηση ε, για την αναχώρα έκθεση, τρεις χώρες από τις παρούς εδώ, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, ήταν αντίθετες. Γιατί οι τάχατες υπάρχουν κάποια εμπιστευτικά δεδομένα εκεί. Ο κύριο Μπερνάρ Μονό για το ΙΕΝΕΦ. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, σα άκουσα προσεκτικά όλου κύριε Υπουργοί και άκουσα ότι θέλετε να καταπολεμήσετε το dumping και την φοροπαπή φυγή στην Ένωση. Και γι' αυτόν τον λόγο υποστηρίζετε τι προτάσει BEPS από τον ΟΑΣΕ υπέροχα. Αλλά 15 χρόνια τα ακούμε αυτά τα λόγια και τα αποτελέσματα δεν έχουν φανεί ακόμα. Και η φοροαποφυγή συνεχίζεται και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με χώρες εκτός, με δυσμενή αντίκτυπο για όλους τους πολίτες. Οι προσπάθειες εναρμόνισης των φορολογικών ε, συστημάτων δεν έχουν προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ε, προωθούν την φορολογική εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσουν τη φοροαποφυγή εταιριών πληροφορικής όπως η Google. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η κατάσταση είναι ότι ο Ευρωπαίος πολίτης εμέσως χρηματοδοτεί μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού θα έπρεπε να κυνηγά την φοροαποφυγή με την ίδια ε, ορμήτη που κυνηγά τι ε, χρηματοδοτήσει από τα κράτη τη. Γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή χωρίς ε, με, όπου όλο και λιγότερο υποχωρεί το κανονιστικό πλαίσιο. Έχουμε μια κατάσταση όπου υπάρχει πλήρης ατιμορρησία των πολυεθνικών εταιριών, των εταιριών συμβούλων και των ε, κρατών και των κυβερνήσεων που εκφεύγουν από το δημοκρατικό έλεγχο και τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω πιο συγκεκριμένα. Θα ε, θέλατε να αναλάβετε ε, μία επιχείρηση συγκεκριμένα ε, εναντίον ε, μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν αξιοποιήσει συστήματα φοροαποφυγής για να ανακτηθούν κεφάλαια και φορολογητέα ύλη. Σας ευχαριστώ. Φτάνουμε λοιπόν στο ΕΛΚ με την Τανούτα Χιούμπνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ, κύριοι Υπουργοί. Θέλω να ασχοληθώ με την ε, αναχώρα έκθεση, αλλά από άλλη οπτική τη διπλή φορολόγηση. Ξέρουμε ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται διεθνώς υφίστανται τον κίνδυνο της διπλής φορολογίας, ιδίως ε, στην περίπτωση του transfer pricing. Η Ένωση για να μειώσει ή να αποφύγει αυτό τον ανεπιθύμητο κίνδυνο ε, διπλής φορολόγησης υιοθετήσαμε τη σύμβαση περί που από ό,τι φαίνεται λειτουργεί, μειώνει τον κίνδυνο διπλής φορολογίας. Εκτός Ένωσης ωστόσο δεν υπάρχουν τέτοιες, τέτοιοι μηχανισμοί ε, δεσμευτικού χαρακτήρα κατά της ε, διπλής φορολογίας. Τώρα ξεκινάει να το συζητά όσα Η πρόκληση λοιπόν στις εκθέσεις αυτές αναχώρα είναι ότι μπορεί να αυξηθεί, να, να αυξηθεί ο ρυθμός των διαφορών για transfer pricing Άρα, μήπω ήταν σκόπιμο να μοιραζόμαστε αυτέ τι αναχώρα πληροφορίε με τι χώρε εκείνε που συμφωνούν να υιοθετήσουν μια διαδικασία ισοδύναμη με αυτή που υιοθετεί η σύμβαση, της, ε, ε Ξέρετε ότι στις ΗΠΑ ε, η αρμόδια επιτροπή του Κογκρέσου έστειλε στο Υπουργείο Οικονομικών μια επιστολή που, ήταν, που έλεγε ότι είναι τελείω αντίθετη με αυτή την αναχώρα έκθεση. Πώς μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο. Είστε έτοιμοι να πείσετε τον υπόλοιπο κόσμο να ακολουθήσει την ίδια πορεία που θέλει να ακολουθήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες η κυρία Μπερές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι εξαιρετικά εξαιρετικό το γεγονό ότι τέσσερις υπουργοί παρευρίθησαν, Γιατί δίνει και ένα σινιάλο το γεγονό ότι παρευρίσκεστε, Ότι όχι μόνο θεωρείται σημαντική την λογοδοσία, αλλά επίσης ότι χωρι εμα χωρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα τα καταφέρουμε. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει διαδικασία της συναπόφασης δεν μπορεί παρά να χρειαστεί και υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θα ήθελα λοιπόν να έχουμε και μια ισότιμη προσέγγιση και να υποστηρίξετε κι εσείς τις προτάσεις του Κοινοβουλίου. Θα, θέλω, θα ήθελα λοιπόν να σας θέσω ερωτήματα πρώτα απ' όλα που, ε, που μου έθεσαν άλλοι οργανισμοί. Όπως για παράδειγμα για μια εταιρεία McDonald's, φαντάζομαι θα την γνωρίζετε, για την οποία γνωρίζουμε ότι εξαιτία της φοροαποφυγής της, από το 2009 μέχρι το 2013, ανέρχεται σε ένα κόστος 10 δισεκατομμύρια ευρώ για τον Ευρωπαίο πολίτη. Ξεκίνησε μια έρευνα στη Γαλλία, επομένως τώρα θα μου πει ο υπουργό ότι δεν μπορεί να μιλήσει γιατί υπάρχει έρευνα να εξελίξει, μάλιστα. Μιας και προχωρά λοιπόν αυτή η, έκθεση, η εξέταση, αυτή η διερεύνηση της υπόθεσης ε, στη Γαλλία, γιατί να μην προσκαλέσουμε τους υπουργούς της Ιταλίας και της Ισπανίας να εξετάσουν τις πρακτικές αυτής της εταιρείας στις δικές τους χώρες. Και αν βρουν κάτι, να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες με τη Γαλλία ω ένα καλό παράδειγμα συνεργασία και πώ μπορούμε καλύτερα να τα καταφέρνουμε όταν εργαζόμαστε από κοινού. Ευχαριστούμε Περβάνς ε, για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον ε, Υπουργό, τον κύριο Παντοάν, το εξή. Κοιτάξτε, την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργό Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα περιστούν τέσσερι φόροι. Ο ένα αφορά την παροχή υπηρεσιών, μετά ε, στην κατοικία, ε, στου αγρότε και ο τέταρτος στις αγροτικές επιχειρήσεις. Ο στόχος λοιπόν είναι βεβαίως να περικοπούν αυτοί οι φόροι. Ε, με τον τρόπο αυτό στόχος είναι να περιοριστεί η φοροαποβηγή. Διότι τελικά αν η κυβέρνηση ανακοινώνει αυτούς τους φόρους, σας είπα ο στόχος είναι να περιοριστεί η φοροαποβηγή. Ίσως θα ήταν λοιπόν σκόπιμο να το έχουμε αυτό κατά νου, κυρίως ε, και σε σχέση με το χρέος η Ευρώπη σε αυτό το τομέα δεν προχώρησε θετικά. Να ρωτήσω το εξής. Εχθές αναφέρθηκε το θέμα της φορολογικής συμφωνίας. Στην Ιταλία η φοροφυγή ανέρχεται σε 21 δις ευρώ. Πολύ ψηλό το ποσό για τον νότο της Ευρώπης προστίθεται η γραφειοκρατία και επίσης και ανυκανότητα ανικανότητα σωστής χρήσης ε, των ε, κρατικών πόρων. Ο νέος λοιπόν, εσείς τι πιστεύετε, θα παραμείνει στο Νότο ή θα θελήσει να φύγει από τον Νότο. Ποια είναι η θα θελησει να φυγει απο το νοτο ποια ειναι η δικη σας γνώμη. Ευχαριστούμε πολύ και τελευταίος ομιλητής για τους σοσιαλδημοκράτες, Ραμόν Χαουρέι. Καλησπέρα και ευχαριστώ. Κύριοι Υπουργοί, μια ερώτηση. Έχει κανεί την εντύπωση ότι, ή μάλλον είμαστε εμεί στην Επιτροπή Τάξη, ότι πραγματικά υπάρχει μια ε, εξέγερση των πολιτών μετά, εν ώψη και της κρίση κατά της φορολογική ε, αποφυγής. Αναφέρθηκαν πράγματα που θεωρούνται ενδιαφέροντα. Πρώτον, την δυνατότητα ενισχυμένων ε, πλειοψηφιών στο ΕΚΟΦΗΝ για λήψη αποφάσεων. Αφετέρου, τη δυνατότητα ενός ελάχιστου ποσοστού φορολόγηση των επιχειρήσεων. Η Επιτροπή ε, όλοι ασχολείται με, τη με την ε, φορολογία των, με, εταιριών που προκύπτει κυρίως μετά το σκάνδαλο του LuxLeaks που επηρεάζει πάρα πολλούς αλλά ο Ισπανός Υπουργός που τον ευχαριστώ που είναι παρός, γιατί ξέρω που είναι παρόν και θέλω να θέσω και δύο σημαντικές ειδικέ ερωτήσεις. Πιστεύετε ότι υπάρχει απάτη και στον ΦΠΑ, ότι υπάρχει δηλαδή μία σημαντική απώλεια διασυνοριακού ΦΠΑ στην Ευρώπη. Δεν είναι αντίστοιχο σκάνδαλο με αυτό των LuxLeaks. Δεν υπάρχουν τεράστιοι διασυνοριακοί τομεί σε μια ενιαία αγορά και μια νομισματική ένωση που, δημιουργία, που, οδηγεί σε μαζική φοροαποφυγή σε έναν βασικό τομέα για εισπράξεων του κράτους. Δεύτερον, μήπως ήρθε η στιγμή να εξετάσει η Ευρώπη το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας φορολογικής υπηρεσίας, μιας εφορίας. Είμαστε σε συνθήκες ε, να πιστεύετε ότι έφτασε η ώρα να υπάρχει μια υπηρεσία φορολογική που θα εισπράττει ή θα παρακολουθεί όλη αυτή τη διαδικασία. Μήπως είναι αναγκαίο να δημιουργήσουμε ένα έμβριο φορολογικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που όλοι τηρήσατε το χρόνο που σας είχα δώσει. Θα πάω και εγώ το λόγο τώρα για να απαντήσω, να θέσω δύο ερωτήσει Στον κύριο Σαπάν και στον Βόλφαγκαν Σόιμπλε. Κύριε Σαπάν, είπατε ότι η εναρμόνιση της φορολογίας των επιχειρήσεων μέσω των ειδικών φόρων κατανάλωσης, των excise duties δηλαδή, είναι κάτι σημαντικό που υποστηρίζει η Γαλλία, αλλά σε ένα 12 μήνο, 18 μήνο χρονικό ορίζοντα. Αυτό με ανησυχεί, γιατί κάποιοι θυμούνται ότι πριν από 20 χρόνια είχε ξεκινήσει η σχετική δουλειά. Τότε ε, ήμουν ε, και υπουργό Οικονομικών, αλλά μετά οι Γάλλοι μέσα στην ε, δημοκρατική φρονημάδα τους ανέτρεψαν την κυβέρνηση και με διώξανε. Αυτό έχει ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια δηλαδή σχεδόν. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας αναδράξουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρία με την υποστήριξη των μέσων και της κοινή γνώμης αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με μια μεγάλη υποστήριξη από πολλά εθνικά κοινοβούλια. Εμεί φέραμε εκπροσώπους όλων των εθνικών κοινοβουλίων εδώ πέρα. Αν δεν αδράξουμε λοιπόν την ευκαιρία θα χαθεί η ευκαιρία αυτή. Και αυτό με οδηγεί σε μια δεύτερη ερώτηση προ τον κύριο Σόιμπλε. Αναμένοντα να υπάρξει κοινός ορισμός του τι είναι φορολογητέο κέρδος, θα περιμένουμε ό,τι μας πει ο κώδικας δεντολογίας. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο της ομάδας ε, κώδικα δεντολογίας και εν συντομία θα έλεγα Υπουργέ ότι η διάγνωση που, στην οποία καταλήξαμε είναι ότι ο κώδικας δεντολογίας είναι μια ωραία κοιμωμένη. Τίποτα δεν γίνεται εκεί πολιτικά. Ακούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον την αποφασιστική βούληση που εκφράσατε παρόντων και με υποστήριξη όλων των συναδέλφων σας εδώ παρόντων να δώσετε και πάλι σημαντικό ρόλο στο, στην ομάδα κώδικα δεντολογίας και να το ανεβάσετε πολιτικά στο επίπεδο που είχε δημιουργηθεί αρχικά. Τώρα είναι διοικητική επιτροπή και αναφέρω. Δεν μπορεί το θέμα αυτό να το κοιτούν μόνο τεχνική. Δίκιο έχετε. Είστε υπέρ του να υποστηρίξετε την πρόταση Juncker εδώ στην Επιτροπή μας την περασμένη εβδομάδα να δημιουργηθεί μια φορολογική επιτροπή αντίστοιχη σε ίδιο επίπεδο με την Νομισματική και Οικονομική Επιτροπή που διαδραματίζει έναν ρόλο που γνωρίζουμε και εκτιμούμε. Κύριοι Υπουργοί, Καλό timing έχουμε. Πέντε λεπτά ο καθένα σα για να απαντήσει. Θέλετε να απαντήσετε με την ίδια τάξη ή με την αντίστροφη. It's up to you. Ο Wolfgang πρώτος και ο Παύλο. Πολύ ωραία αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητέ Αλά. Θα ήθελα να ξεκινήσω απαντώντας την ερώτηση του Πρόεδρου, στη, την τελευταία ερώτηση. Ξεκινάω με αυτήν και θα ε, προσπαθήσω να απαντήσω και όλες άλλες πολλές ερωτήσεις που μου ετέθησαν. Εγώ λοιπόν είπα ότι αυτή η ομάδα του κώδικα δεοντολογίας ε, πρέπει να στηριχθεί γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση για να προχωρήσουμε. Όμως ε, πρέπει να σας πω ότι στηρίζω και αυτό που είπε ο κύριος Γιούνκερ, δηλαδή να προχωρήσουμε ακόμα ένα βήμα πιο πέρα. Με μια λέξη λοιπόν θα έλεγα ότι σαφώς η απάντηση είναι ναι. Ε, προς την κυρία ε, Φερέρα. Γιατί μέχρι τώρα, ρώτησε η κυρία Φερέρα, δεν ασχοληθήκατε. Ίσως ε, να θυμάστε το μπροκάτοχό μου ε, στη Γερμανία, τον Υπουργό Οικονομικών, ε, που ήθελε να στείλει το υπηκό στο Λουξεμβούργο και η απάντηση του Λουξεμβούργου Υπουργού ήταν, ξέρετε, καλά, έχουν έρθει οι Γερμανοί μια φορά στο Λουξεμβούργο, καλό είναι να πάνε να μείνουν εκεί που είναι, δεν χρειάζεται να ξανάρθουν. Γιατί το λέω αυτό, για να πω ότι υπάρχουν προβλήματα συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν τα όρια, υπάρχουν τα σύνορα. Και εκτός αυτού αυτές τις μορφές tax rulings δεν τις είχαμε μέχρι σήμερα. Σήμερα έχουμε τους ε, διεθνείς ορισμούς που δίδουν έτσι μια ευρύτερη ερμηνεία στα tax rulings, φορολογικές αποφάσεις. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας πω ότι εμείς υποβάλαμε όλες τις ερωτήσεις ε, στην Επιτροπή, δώσαμε όλες τις απαντήσεις. Εκείνο που θα μου επιτρέψετε να προσθέσω είναι ότι όλοι μας παρεπιπτόντος ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τώρα μπορεί να σας αρέσει, μπορεί να μην σας αρέσει, εγώ όμως είμαι πολλά χρόνια κοινοβουλευτικός ε, για να ξέρω και προσέξτε θα έλεγα μην έρθετε σε ανταγωνισμό μαζί μου όσον αφορά τουλάχιστον τα κοινοβουλευτικά μου χρόνια. Επανέρχομαι Έρχομαι λοιπόν και να λέω ότι οι κανόνες δεν εφαρμόζονται πάντα και δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν γιατί ξέρετε δεν υπάρχουν οι αρμοδιότητες που νομίζει κανείς ότι έχει. Ας πούμε στην Ευρώπη δεσμευόμεθα από το πρωτογενές δίκαιο, το δίκαιο των συνθήκων. Γνωρίζω ότι στη Γερμανία οποτεδήποτε ε, εκδώσω μια απόφαση μου λένε ξέρετε κάτι τα παρέμει και το κοινοβούλιο θα εμπερδευτούν τα πράγματα άρα δηλαδή για να μην υπάρχουν δυσκολίες τηρούμε το πρωτογενέ δίκαιο. Αυτή είναι η κατάσταση. Κατά τα άλλα, στη Γερμανία είμαι υποχρεωμένο να τηρώ το γερμανικό σύνταγμα και άλλε χώρε το δικό του σύνταγμα. Και να σα πω κάτι, στη Γερμανία η φορολογική διαχείριση εμπίπτει στι αρμοδιότητε των κρατηδίων. Η, ε, Σύμμαχοι το 49 αποφάσισαν να φτιάξουν τα κρατήδια και γιατί, γιατί είχαμε αυτό το μοιραίο παρελθόν Τότε λοιπόν μας επέβαλα να έχουμε αυτή τη μορφή διακυβέρνησης ως εκ τούτου δεν είναι ενιαία φορολογική διαχείριση. Ξέρετε αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον Υπουργό Οικονομικών αλλά να μην σας τα εξηγήσω τώρα. Τώρα όσον αφορά τις ε, αναχώρα εκθέσεις ξέρετε κάτι εξαρτώμε από το να συμφωνούν και τα κρατήδια σε μένα που πολλές φορές δεν, κρα... δεν συμφωνούν και στη Γερμανία, μόνον αυτό αλλά έχω και τη δεύτερη βουλή που και αυτοί μου δημιουργούν τεράστια προβλήματα, μεγαλύτερα από ό,τι σε εσά. Τέλο πάντων, εγώ δεν ήρθα εδώ σήμερα για να μυρολογώ και να γκρινιάζω. Απλά να σα πω γιατί χρειάζεται χρόνο και πού βρίσκονται οι αντιδράσει. Συνάδελφε κύριε Τόιρ, να σα πω το εξή. Το έχετε πει επανειλημμένα και δεν καταλαβαίνω την ε, έλλειψη υπομονή που επιδεικνύεται. Από την άλλη, μην ξεχνάτε ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουμε όχι μόνο τη φοροδιαφυγή, αλλά και και το περιορισμό του περιθωρίου διαφορετικών νομοθετικών και φορολογικών ρυθμίσεων. Έχουμε προχωρήσει πολύ περισσότερο από ό,τι πίστευε κανείς μέχρι πριν από πέντε χρόνια. Τώρα το θέμα είναι κατά πόσον λόγω της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα. Ας πούμε θα πρέπει να ασχοληθούμε με την ψηφιοποίηση φορολογικών ρυθμίσεων και πολλά άλλα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι θα πρέπει κανείς να αναζητήσει πολύ σοβαρά λύσεις. Πριν από κάποια χρόνια ούτε να το σκεφτούμε δεν θα τολμούσαμε ότι θα υπήρχε η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, και από το 17, 1η Ιανουαρίου του 17 θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Αυτό λοιπόν είναι ένα βήμα που πάρα πολλά κράτη δεν μπορούσαν καν να το φανταστούν. Στη Γερμανία εξάλλου υπάρχει και το φορολογικό απόρριτο. Αυτός είναι ένας από τους λόγους γιατί συνάδελφε Λούκε τα κρατήδια δίνουν κάποιες πληροφορίες και άλλες πάλι όχι. Γιατί ξέρετε κάτι, το φορολογικό απόρριτο είναι εδώ και πάνω από 100 χρόνια βασική αρχή των αρμοδιοτήτων και της φορολογίας ε, στη Γερμανία, φορολογία των ε, κρατηδίων στους φορολογούμενους λέει κανείς ότι θα πρέπει να αποκαλυφθείτε για να γίνεται η σωστή φορολογία και εκεί όμως όπως σας είπα λόγω διαφορετικών αρμοδιοτήτων υπάρχουν κάποια όρια. Τώρα όσον αφορά τη φορολογική βάση ε, φόρου επί των επιχειρήσεων γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν διαφορές ε, στα διάφορα κρατήρια, πολύ μεγάλες διαφορές άρα δηλαδή το εγχείρημα είναι φιλόδοξο. Εγώ όμως θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε με ενθουσιασμό και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπή βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Ένα άλλο ερώτημα. Αν έχουμε υπολογίσει ποια είναι τα ποσά τα οποία διαφεύγουν από τα δημόσια ταμεία λόγω της ε, φοροδιαφυγής. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν μπορεί κανείς όλα αυτά να τα συνδέσει με κοινοβουλευτικές ε, απαντήσεις. Έχουμε κάνει τους υπολογισμούς μας, αλλά δεν θα απαντήσουμε ποτέ σε τέτοια ερώτηση. Σε εθνικό επίπεδο προσπαθούμε Προσπαθούμε στο βαθμό του δυνατού να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή, αλλά ξέρετε κάτι, αυτό ε, είναι ένα ερώτημα που αφορά και πάλι τη συνεργασία με τα κρατήδια στη Γερμανία, το θέμα των BEPS. Εμείς το ξεκινήσαμε, μόνο εμείς, μόνο που θα πρέπει να εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό δίκαιο και τα πράγματα θα προχωρήσουν ε, γρήγορα ή όχι, ανάλογα με το πώς θα προχωρήσουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Ζητώ συγγνώμη κύριοι και κυρίες που ξεπέρασα το χρόνο μου. Ευχαριστώ. Ο Λουίς έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τις προάλλες στο άτυπο Κουφίν που είχαμε στο Λουξεμβούργο υπό την προεδρία του Λουξεμβούργου έκανα μια σκέψη, το είπα, ότι αν μου λέγανε ότι θα είχαμε πριν από λίγα χρόνια ένα άτυπο εκοφήν με Λουξεμβούργο πρόεδρο και θα συζητούσαμε την, ε, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροποφυγής, θα είχα γελάσει. Αυτό έγινε πραγματικότητα ωστόσο και αυτό δείχνει ότι αλλάζει η κατάσταση, αλλάζουν οι καιροί και προς το καλύτερο θα έλεγα. Δεύτερον, τέθηκαν μια σειρά ερωτημάτων, θεμάτων πιο ειδικών και για την Ισπανία για την αναχώρα ενημέρωση. Εμείς το εγκρίναμε και το εφαρμόζουμε με ένα, χρόνο, ένα χρόνο σε σχέση με αυτό που προέβλεπε ο ΩΣΑ. Πιστεύουμε ότι είναι ένα βασικό βήμα. Πάντα πιστεύαμε ότι η, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ήταν θετική και αυτό το είχαμε προτείνει με τη Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία και Ιταλία και γίνεται. Και υπάρχει μια επίπτωση δικτύου. Όσο περισσότερες χώρες είμαστε, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η ανταλλαγή πληροφοριών. Για το Γιβραλτάρ τώρα. Είναι μια σπαζοκεφαλιά για τις ε, φορολογικέ αρχές της Ισπανία, μόνιμη σπαζοκεφαλιά το φορολογικό σύστημα εκεί. Διότι το φορολογικό καθεστώς ε, του Γιβραλτάρ πάσχει από έλλειψη διαφάνειας, είναι εξαιρετικά αδιαφανές και η βασική φορολογική υπηρεσία που υφίσταται τις επιπτώσεις είναι ακριβώς τη ισπανική. Το Γιβραλτάρ έχει πολύ χαμηλή φορολογία και ταυτόχρονα μία ακατάλληλη και πολύ, συχνή, πολύ συχνά ε, λάθος χρησιμοποίηση των tax rulings. Οι ισπανικές φορολογικές αρχές θεωρούν ότι ε, δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο στο σχέδιο έκθεση ενώ παραμένουν οι ανοιχτέ ε, υποθέσει κατά άλλων κρατών μελών. Δεν περιλαμβάνεται τίποτα στην έκθεση. Ποιο είναι ο λόγο τον οποίο στο σχέδιο έκθεση δεν αναφέρονται ζητήματα που επιπλέον η ίδια η Επιτροπή σε ανάλυση κρατικών ενισχύσεων θεωρήσε ότι υπήρχαν 165 περιπτώσεις νομίζω που είχε κρίνει ότι ήταν τα tax rulings αυτά ήταν παραβίαση της νομοθεσίας για, την κρατική, κρατικές ενισχύσεις, κάτι σημαντικό νομίζω. Έγινε και μία μνήα στο θέμα της διαφάνειας. Η Ισπανική κυβέρνηση υποστηρίζει το πακέτο διαφάνειας που υπέβαλε η Κομισιόν για τα θέματα φορολογικής ε, ε, πολιτικής. Υποστηρίζουμε, υποστηρίξαμε την οδηγία για την διοικητική συνεργασία και είμαστε πρωτοπόροι, όπω είπα, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Λογικά, στο πλαίσιο των φορολογικών μεταρρυθμίσεων, υιοθετήσαμε πολλά μέτρα προ όφελο τη διαφάνεια. Έλεγα προηγουμένως για την αλλαγή που έγινε στην νομοθεσία σε ό,τι αφορά την ευθύνη των ε, ε, διοικητικών συμβουλίων, ε, σε επιχειρήσεων, σε παράνομες συμπεριφορές επιχειρήσεων ή την αποκάλυψη των ε, καταδικαστικών αποφάσεων. Η διαφάνεια προφανώς πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα που δείχνουν ε, αποφασιστικότητα και ταυτόχρονα προστασία και των δεδομένων. Σε ό,τι αφορά άλλες πιθανές, ε, το, άλλους πιθανούς τομείς ε, προόδου αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής σε άλλους τομείς φορολογίας δεν είναι κακή ιδέα. Υπάρχουν μηνύματα ότι μπορεί να γίνονται κάτι τέτοιο, όχι μόνο για τον, τη φορολογία των επιχειρήσεων και για το ΦΠΑ συμφωνώ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε κάποια βήματα Τώρα για την Ευρωπαϊκή Φορολογική Υπηρεσία, εγώ είμαι φιλοευρωπαίος πάντα, αλλά νομίζω ότι πριν γίνουν κάποια βήματα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, ξέρετε ότι μερικές φορές ε, το καλύτερο είναι εχθρό του καλού. Σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν πολύ πιο σημαντικό να εφαρμόσουμε τις να εγκρίνουμε και να εφαρμόσουμε τις εκκρεμίες οδηγίες, να υιοθετήσουμε ό,τι έχει να κάνει με τα BEPS, σαν ένα minimum standard σε όλη την Ένωση και μετά να δούμε άλλες εξελίξεις. Κάποιο σχόλιο εκτός μικροφώνου γίνεται. Εκτός μικροφώνου κάποιες παρατηρήσεις. Α, τα McDonald. Δεν τα ξέρω τα, την ιστορία των McDonald. Μα δεν σας αρέσουν τα McDonald. Ο Μισελ Σαμπρά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που μου απευθύνατε. Καλύτερα δεν θα ήταν πιο γρήγορα και πιο δυνατά και καλύτερα για όλα τα θέματα θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε τις εξελίξεις και την πρόοδο που έχει συμμετοχθεί τα τελευταία χρόνια. Σε διεθνές επίπεδο κυρίως, στο επίπεδο των G20, που θα έλεγα ότι είναι και το πιο σημαντικό επίπεδο, αν μιλάμε για την βελτίωση της φορολογίας επιχειρήσεων. Γιατί δεν είναι το ζήτημα να εναρμονίσουμε μόνο τα ευρωπαϊκά φορολογικά συστήματα, αλλά να δούμε και τι θα κάνουμε με τους φορολογικούς παραδείσους. Όταν βλέπω πώς περάσαμε σε τρία χρόνια και τι θα πρόκειται να συζητήσουμε στην Αντάλια τώρα, έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο. Γιατί πολλοί συνάδελφοι, πολλοί από εσά το αναφέρατε ότι για τα ζητήματα αυτά το συζητάμε επί χρόνια. Τώρα πια έχουμε φτάσει στο σημείο που μπορούν να λεφθούν και αποφάσει. Καταλαβαίνω την ανυπομονησία, αλλά ε, τα τελευταία τρία χρόνια νομίζω ότι έχουν επιταχυνθεί πολύ οι εξελιξει. Κάτι ακόμα. Πρέπει να υπάρχει μια ιεράρχηση τη προτεραιότητα των διαφόρων ζητημάτων. Είναι ένα ζήτημα η φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη. Εδώ πρέπει να λάβουμε αποφάσεις ο καθένας στη χώρα του. Είναι ένα θέμα στο οποίο η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στο οποίο έχει ε, δραστηριοποιηθεί εναργά η Γαλλία, ιδιαίτερα στο θέμα του ΦΠΑ. Και επίσης εκεί χρειάζεται μια καλή ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο, δηλαδή φορολογικών στοιχείων και για φυσικά και νομικά πρόσωπα, Εκεί έχουν επίσης γίνει μεγάλη ε, πρόοδοι. Το διαπιστώνω κοιτώντα τα φορολογικά έσοδα από Γάλλους πολίτες που είχαν και έχουν λογαριασμού στο εξωτερικό. Όχι μόνο κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και κράτη εκτός Ένωσης και βλέπω ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Γιατί, Γιατί αποφασίσαμε ε, μεταξύ μας οι χώρες της Ένωσης να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Κάτι ακόμα, το επόμενο μάλλον στάδιο, είναι η καταπολέμηση του ε, φορολογικού προγραμματισμού όταν αυτός είναι ε, Που είναι και το σημαντικότερο ζήτημα που αφορά αυτήν εδώ την Επιτροπή. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε βήματα, αλλά πρέπει αυτά να είναι μεθοδικά. Γιατί πολλά επιμέρους ζητήματα και πολλές ε, διαφορετικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται για αυτό τον αθέμητο ε, φορολογικό προγραμματισμό. Και σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει επιτάπητος μια οδηγία την οποία η Γαλλία και άλλες χώρες θα θέλαμε να υιοθετηθεί, να εγκριθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς για να μην ξαναδούμε τα φαινόμενα του παρελθόντος να παραλαμβάνονται. Μετά, τρίτο στάδιο, είναι η εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων. Επίσης πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί βεβαίως μπορούμε να δεχτούμε μια, ένα φορολογικό ανταγωνισμό όταν αυτός βρίσκεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε τις πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μας. Γιατί στην πραγματικότητα, αν τους επιτρέψουμε αυτές τις μεγάλες διαφορές, θέτουμε τις χώρες μας να ανταγωνίζονται μία στην άλλη. Την άλλη. Και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε, θα οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα για κράτη-μέλη της Ένωσης. Επίσης, έχουμε το, το ζήτημα μιας συζήτησης που κρατάει εδώ και πολύ καιρό, της λήψης αποφάσεων και για το, της διακυβέρνησης. Μέχρι στιγμής έχουμε το σύστημα της α, ε, ομοφωνίας. Και κατά την άποψή μου πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, πρέπει να τροποποιήσουμε τις συνθήκες που μας περιορίζουν αυτή τη στιγμή έτσι ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις και με, και με ενισχυμένη πλειοψηφία στα ζητήματα τα φορολογικά, όχι μόνο ε, με την ε, ομοφωνία που γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματά της. Γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματά της στο επίπεδο του Eurogroup, φανταστείτε ποια είναι στο σύνολο των κρατών της Ένωσης. Επίσης, θέλω να απαντήσω σε ερωτήματα που απευθύνθηκαν συγκεκριμένα στη Γαλλία για το ζήτημα της έρευνας και της ανάπτυξης και το ειδικό φορολογικό ε, καθεστώς. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο έχουμε δημιουργήσει στη Γαλλία, Credit δηλαδή μια δυνατότητα χρηματοδότησης, έμεσης χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που σκοπεύουν να κάνουν προγράμματα έρευνας και αυτό είναι πλήρως διαφανές. Δεν κρύβεται τίποτα. Είναι δημοσιο, δημόσια αυτά τα στοιχεία. Εξάλλου, ε, εμεί προσπαθούμε, εισάγουμε αυτά τα μέτρα γνωρίζοντα ότι η φορολόγηση των επιχειρήσεων στη Γαλλία είναι υψηλή σχετικά. Ε, φτάνει μέχρι 38% στις, ε, στις, για ορισμένα είδη επιχειρήσεων, ενώ ο μέσος όρος, στην Ευρώπη είναι περίπου 28%. Επομένως, αυτό το σύστημα της έμεσης ε, φορο, ε, φορολογικών κινήτρων, φορολογικών ελαφρύνσεων για την έρευνα, δεν ε, είναι μέθοδος φοροφυγής, αντιθέτως είναι ένα διαφανές σύστημα για να ενισχύσουμε την έρευνα. Σας ευχαριστώ, ελπίζω να απάντησα και στα συγκεκριμένα και στα γενικότερα ερωτήματα. Ε, ε δεν θα μιλήσω καν για τα McDonald's γιατί είναι ακριβώς το αντίθετο της γαλλικής κουβιζίνα και δεν μου αρέσουν καθόλου. Αλλά, όχι, θα σα απαντήσω λίγο. Σε πολλά θέματα από αυτά που δημοσιοποίησαν τα LuxLeaks. Η γαλλική δημόσια προσπαθεί, αφού κάνει την απαραίτητη απεξεργασία των στοιχείων, να ζητήσει από τις επιχειρήσεις που είχαν φόρο αποφύγει να πληρώσουν το φόρο που τους αναλογεί. Και την περασμένη εβδομάδα άλλωστε η κυρία Φεστάγκη είχε πει ότι θα ξεκινούσε πολύ περισσότερες έρευνες για κρατικές ενισχύσεις από ό,τι πίστευε στην αρχή. Ας ε, χειροκροτήσουμε και τον κύριο Σαπάν γιατί είχατε χειροκροτήσει και τους άλλους. Πριν δώσω το λόγο για να κλείσει τον κύριο Παντοάν. Τέτοια ώρα που είναι να μην σας φάω πολύ χρόνο. Δύο γενικά θέματα. Τα είπαν και οι συνάδελφοι όλοι λένε τι κρίμα που είναι η μικρή πρόοδος. Αν δείτε πριν από λίγα χρόνια στο ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης θα δείτε ότι η πρόοδος ήταν τεράστια. Το να μιλάμε για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, για να μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι το τραπεζικό απόρριτο δεν υπάρχει πια, ήταν κάτι αδιανόητο πριν λίγα χρόνια. Ήταν μία από τις λίγες θετικές απαντήσεις στην μεγάλη κρίση. Η δυνατότητα να λέμε ότι σήμερα πρέπει να εξετάσουμε όχι τόσο τη διπλή φορολόγηση, αλλά να αποφύγουμε την διπλή μη φορολόγηση, είναι ένα άλλο μήνυμα του ότι προχωρούμε προς μία θεσμική αρχιτεκτονική της Ένωσης με κοινούς κανόνες για τα κράτη-μέλη της Ένωσης που θα εξασφαλίζουν ένα level playing field και ταυτόχρονα θα αποφεύγει την, τον αθέμητο ανταγωνισμό. Έχω την άποψη λοιπόν ότι στην πράξη έγινε μεγάλη πρόοδος. Βεβαίω πάντα υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν και αυτό αποτελεί κομμάτι της ε, θεματολογίας για τα μπέψε. Για τη φορολογική εναρμόνιση. Είπε ο Μισελ κάποια πράγματα. Η φορολογική εναρμόνιση είναι ένα σύνθετο ζήτημα στην Ευρώπη Ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι πρέπει να εναρμονίσουμε και τι πρέπει να αφήσουμε στον ανοιχτό και διάφανο ανταγωνισμό. Σίγουρα οι κανόνες για μια κοινή φορολογική βάση ε, είναι ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση μιας ε, ισότιμης αντιμετώπισης των επιχειρήσεων. Για την Ιταλία κάποιες απαντήσεις. Πρώτον, δεν είναι αληθές, δεν είναι αληθές όσο είμαι εγώ τουλάχιστον ότι, ότι η χώρα αντιτίθεται, αντιτάχθηκε στο country by country report στο ECOFIN. Αν έχετε τέτοιες ε, διαρροέ είναι λάθος. Ε, βρείτε άλλους πληροφοριοδότες. Δεύτερον, τι κάνει η Ιταλία στις ε, διαθροντικές μεταρρυθμίσεις που έχει υιοθετήσει ε, η Ιταλία έχει εισάγει και ένα νόμο πλαίσιο για τη φορολογία στην ουσία. Κάποιοι από τους κανόνες που έχουν να κάνουν με, τον, ε, με την υλοποίηση αυτή του νόμου πλαισίου έχουν και την μείωση της ε, κατάχρησης που υπήρχε και την υιοθέτησε το country by country report Κάνει λοιπόν ό,τι μπορεί η χώρα για να εκμεταλλευτεί το νέο κλίμα φορολογικής διαφάνειας και να συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός πιο δίκαιου και διάφανου φορολογικού, ενιαίου φορολογικού πλαισίου όπου θα μπορούσε να υπάρχει μια fair competition. Να απαντήσω στην κυρία Ματουτσέλο ότι δεν συμφωνώ με την ιδέα ότι η αναγγελία περικοπών φόρων είναι κίνητρα στην φοροδιαφυγή. Το αντίθετο πιστεύω. Όταν αναγγέλουμε ότι περικόπτουμε φόρους, το κίνητρο για τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή μειώνεται και επιτρέπει να υπάρχουν τελικά έσοδα στον δημόσιο κορβανά και να βελτιωθεί η φορολογική ε, δικαιοσύνη. Σας δίνω και ένα λεπτό από τα πέντε που είχα. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι εκτιμήσαμε όλοι αυτά που μας είπατε. Να πω δύο λόγια για τα φορολογητέα κέρδη. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος ποιος είναι. Πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό που θέλουμε εδώ είναι να μπορούν να φορολογούνται τα κέρδη ούτως ώστε αυτά που υπέφεραν οι προκάτοχοί μας για τον ΦΠΑ πριν από 40 χρόνια. Και οι Βρετανοί φίλοι δεν είχαν αντιταχθεί τότε σε αυτό, δεν είχαν πει ότι αυτό προσβάλλει την εθνική κυριαρχία. Ο φορολογικός ανταγωνισμός είναι ένα αντικειμενικό δεδομένο που δεν μπορούμε να χτυπήσουμε. Κάποιοι από εμά το θεωρούν υγιές. Yes. Αντίθετα, κανένας καλόπιστος άνθρωπος δεν μπορεί να αρνηθεί ότι στον φορολογικό ανταγωνισμό θα πρέπει να εφαρμόζουμε τους κανόνες και τις αρχές που εφαρμόζονται σε όλους τους άλλους τομείς. Διαφάνεια, νομιμοφροσύνη, δικαιοσύνη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή ο φορολογικός ανταγωνισμός γίνεται ε, σε, στο σκοτάδι με ψέματα και με αδικίες. Αυτό δεν μπορεί να το δεχθεί κανένας. Εμείς θεωρούμε εξαιρετικά θετικό το ότι οι υπουργοί που είναι εδώ παρόντες σήμερα και που εκπροσωπούν τις δυνατότερες ε, οικονομίες της Ευρωζώνης τουλάχιστον είναι υπέρ αυτής της θεμελιώδους μεταρρυθμίσεως. Θα τους εκλυπαρούσα εσείς εκπρόσωποι των μεγάλων χωρών μη φοβάστε τις μικρές. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου, τέλος συνεδριάσεως.